All right, thank you very much. Um, I would start by uh, having uh, an Θα κάνω πρώτα ανακοινώσεις. Ο κύριος Μπροκ, πρόεδρος μας, είχε άλλη ανηλυμένη υποχρέωση με την Ουκρανία και γι' αυτό δεν θα έρθει. Δεν θα έρθει. Πρώτο θέμα για σήμερα είναι η συνάντησή μας με... με... Α, ναι, ευχαριστώ. Έχω ένα θέμα με την απουσία του κυρίου Μπροκ. Έχει ιδιωτική συνάντηση με τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης στην Ουκρανία. Αλλά και συνοδεύει, αντιπροσωπεύει έτσι την καγκελάριο. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η συνάντηση. Κοιτάξτε, δεν είναι ερώτηση αυτό, ούτε το γράφει εδώ πέρα, οπότε όχι να ζητήσετε από τη γραμματεία να συμπληρώσει αυτή την πληροφόρηση. Γιατί θα θέλαμε να πετύχει η αποστολή του κυρίου Μπαροκ. Μάλιστα. Θα διαβάσω τώρα αυτά που έχω μπροστά μου, θα διαβάσω. Τον περασμένο Δεκέμβριο ψηφίσαμε το καινούργιο εξωτερικό εργαλείο ε, χρηματοδότησης και οι νομομαθείς μας τελικά μπόρεσαν να ελέγξουν τα πράγματα μόνο μετά την ψηφοφορία. Η γραμματεία σας έχει μοιράσει τα κείμενα που διόρθωσε η νομική υπηρεσία. Βέβαια οι αλλαγές αυτές δεν αλλάζουν καθόλου την ουσία της συμφωνίας που επετεύχθη στον τριμερή διάλογο, απλώς γλωσσικά και νομικά συμμορφώθηκε. Η γραμματεία της επέξα φρόντισε να, τα δεχτούν, να δεχτούν τις αλλαγές αυτές και όλοι οι συντονιστές. Αν δεν έχετε λοιπόν αντιρρήσεις, αυτή η νέα μορφή θα εγκριθεί και θα σταλεί στην Ολομέλεια. Τώρα έχουμε όπως σας έλεγα την ευχαρίστηση να έχουμε μαζί μας τον κύριο Ίγκορ Κόρμαν, εκπρόσωπο του Κοινοβουλίου της Μολδαβίας, πρόεδρο, που θα μας μιλήσει για τις σχέσεις ΕΕ Μολδαβίας μετά από τη διάσκεψη κορυφής του Βίλνιους. Ορίστε κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πάσχου. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ και μέλη της ΕΠΕΞ, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή η παρουσία μου εδώ σήμερα μπροστά στην Επιτροπή Εξωτερικών στα πλαίσια της επικείμενης λήψης αποφάσεων που αφορούν τη Μολδαβία και το μέλλον της. Από το 2009 η προτεραιότητα της Μολδαβίας ε, στα εξωτερικά ήταν η ευρωπαϊκή προτεραιότητα. Η χώρα μας άρχισε διαπραγματεύσεις με την Ένωση Σύνδεσης και για το CFTA και για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Αναλάβαμε τη δέσμευση να εφαρμόσουμε ό,τι ίσχυε στην νομοθεσία για το σεβασμό των ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων ως βάση της σχέσης μας με την Ένωση. Και έχουμε αρχίσει στεναρές νομικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις για θέματα συνόρων και μετανάστευσης, δημόσιας τάξης, δικαιοσύνης που εφαρμόζεται σε συνδυασμό με συμμετοχή με την Ένωση καταπολέμηση της διαφθοράς επίσης καθώς και η περιφερειακή συνοχή και η λογοδοσία για δικαστές. Και το νέο ποινικό δίκαιό μας προβλέπει και εκτεταμένες κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων. Έχουμε προβλέψει επίσης ενδυνάμωση των μηχανισμών προστασίας γιατί πιστεύουμε ότι έτσι θα καλλιεργηθεί και στη Μολδαβία ένας πολιτισμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δίκαιας κοινωνίας. <clears throat> Αυτές και άλλες μεταρρυθμίσεις είχαν βέβαια και κάποιο χρηματικό και κοινωνικό κόστος. Οι νέες χώρες μέλη της Ένωσης θα συμφωνούσαν ότι το ταξίδι προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν είναι εύκολο. Η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση στη Μολδαβία αντιμετώπισε πολλές προκλήσεις όπως πολιτική αστάθεια, έλλειψη εμπειρίας στη διακυβέρνηση, και την απουσία επικοδομητικού διαλόγου με την αντιπολίτευση καθώς και οικονομικά προβλήματα σε εκείνη την δύσκολη περιοχή. Πολλές από αυτές τις προκλήσεις παραμένουν. Αλλά και αυτές οι προκλήσεις και άλλες δεν μας αποθάρρυναν διότι πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος. Γιατί οι ευρωπαϊκές αξίες που συμμεριζόμαστε και εμείς είναι εκείνες που μας βοήθησαν και τον ε, φιλοευρωπαϊκό συνασπισμό που είναι στην κυβέρνηση να συνεχίσουμε τον εξυγχρονισμό της Μολδαβίας. Η συμφωνία σύνδεσης πέρυσι ήταν ένα σημάδι, ένα σημείο της πρόοδου που έχει επιτύχει η Μολδαβία Επίσης εφαρμόσαμε όλες τις διατάξεις που προέβλεπε το σχέδιο δράσης για την απελευθέρωση των θεωρήσεων και το αναγνώρισε λίγες μέρες πριν τη διάσκεψη του Βίλνιους η Κομισιόν προτείνοντας να καταργηθούν οι θεωρήσεις για τους πολίτες της Μολδαβίας. Ευχαριστώ για αυτό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βοήθειά της και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξη που έκανε αυτές τις μεταρρυθμίσεις δυνατές σε εποχή μάλιστα που η Ένωση αντιμετώπιζε ταυτόχρονα δικές της εσωτερικές προκλήσεις. Αγαπητοί συνάδελφοι, φέτος, δηλαδή το 2014, είναι ζωτικό έτος για τη χώρα μας. Θα δούμε τα αποτελέσματα που είχαν όλες οι φιλοευρωπαϊκές μας προσπάθειες. Στο τέλος, στις εκλογές δηλαδή, οι πολίτες θα κρίνουν αυτές οι εξυγχρονιστικές μεταρρυθμίσεις κορυφώνονται με αυτή την κατάργηση των θεωρήσεων. Η αναγνώριση οφείλεται στο... φαίνεται και από τις προσπάθειες άλλων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης όπου η απελευθέρωση των θεωρήσεων σήμανε τον δρόμο της ε, Ένωσης για τη φέρνει και τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή οικογένεια εδώ. Ευχαριστώ την ΕΠΕΞ και την ΛΥΜΠΕ γιατί αναγνώρισαν ότι η Μολδαβία πληρούσε όλα τα κριτήρια για την απελευθέρωση των θεωρήσεων και τη διακίνηση Μολδαβών στην Ένωση. Επίσης πρέπει να συνεργαστούμε με ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ προσβλέπουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να καταλήξουμε σε τελικό, τελειωτικό και θετικό αποτέλεσμα. Το άμεσο μέλλον για τη Μολδαβία σημαίνει επίσης και την έγκριση και επικύρωση της Συμφωνίας Σύνθεσης και του CFTA. Πριν από τις εθνικές εκλογές τον Νοέμβριο. Πέρα όμως από τις θεωρήσεις και την προετοιμασία για την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνθεσης χρειάζεται να γίνουν και άλλα πολλά. Θα συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις μας. Πριν υπογραφεί η Συμφωνία Σύνδεσης και αφού εγκριθεί το πρόγραμμα που προβλέπει η Ένωση, θα σχεδιάσουμε ένα διεθνές πρόγραμμα δράσης για την επικύρωση. και θα διαδώσουμε τα ωφέλη που έχει για τη Μολδαβία η σύνδεση ώστε να υπάρχει επικοδομητικός και χρήσιμος εθνικός διάλογος με όλους τους πολίτες μας. Τα ωφέλη από την ολοκλήρωση στην Ένωση, όπως φαίνεται και από το CFTA, την απελευθέρωση των θεωρήσεων και τη Συμφωνία Σύνδεσης, θα καταλήξουν σε απτά υλικά ωφέλη για τους πολίτες. που θα καταπολεμήσουν την πολιτική και οικονομική μας απομόνωση. Χρειάζονται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να βρεθούν βιώσιμες λύσεις για όλα αυτά τα προβλήματα. Ε, θα ήθελα να τονίσω εδώ την στεναρή πολιτική υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καταδίκασε αυτόν τον μήνα την παραβίαση των δικαιωμάτων παιδιών στα παρασχολικά προγράμματα στην υπερθενιστερία. Εκτιμούμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσφατα έδειξε ότι ευαισθητοποιείται για τα προβλήματα της Μολδαβίας απελευθερώνοντας και την εισαγωγή μολδαβικών ίνων στην Ένωση. Τέτοια αλληλεγγύη είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί η αγορά της Ρωσικής Ομοσπονδίας δυστυχώς είναι κλειστή για μας. Πρέπει να έχουμε την ίδια ενωσιακή προσέγγιση και για άλλα προϊόντα όπως φρούτα και λαχανικά για να βοηθηθεί η γεωργία μας και η μετα... ο μεταποιητικός τομέας για να γίνει ανταγωνιστικότερος. Και έρχομαι τώρα στο θέμα της οικονομικής και των οικονομικών και πολιτικών σχέσεων με τους παραδοσιακούς ανατολικούς μας εταίρους. Όπως κάθε ανεξάρτητο κράτος και η Μολδαβία είναι υπεύθυνη για τη λήψη αποφάσεων που να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των πολιτών της. Και γι' αυτό αποφασίσαμε να συνεχίσουμε την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού προτύπου. Δεν είναι γεωπολιτική επιλογή, αλλά επιλογή εξυγχρονισμού. Και δεν θα έπρεπε να αντιταχθεί στις σχέσεις που έχουμε τώρα με χώρες της CIS, της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών. Αγαπητοί φίλοι, είμαστε στα πρόθυρα της βελτίωσης των σχέσεών μας με την Ένωση. Παρά την ύπαρξη δυνάμεων που είναι κατά της ευρωπαϊκής προοπτικής της Μολδαβίας, ο κυβερνητικός συνασπισμός είναι αποφασισμένος να διασφαλίσει πολιτική σταθερότητα και ευρωπαϊκή οδό. Για μας δεν υπάρχει επαναχώρηση στο τρέχον γεωπολιτικό περιβάλλον θα θέλαμε να μπορέσουμε να υποφεληθούμε από τη συνεχή στήριξη των φίλων μας στην Ευρώπη, ώστε η Μολδαβία να γίνει πραγματικά ευρωπαϊκή χώρα. Σας κατευχαριστώ για την υποστήριξή σας και γιατί μου δώσατε τη δυνατότητα να συμμεριστώ τις σκέψεις μου μαζί σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Είστε αποφασισμένος και εσείς και η χώρα σας και πραγματικά αυτά θέλουμε να ακούμε στις Βρυξέλλες από εσά γιατί επενδύουμε στη χώρα σας και θα θέλαμε να δούμε να συνεχίζουν την προσήλωσή τους ε, στην οδό που έχει ακολουθηθεί. Σε σχέση με το θέμα του ίνου, θυμάμαι ένα πρώην παίκτη χόκεϊ που είχε πει ότι αν θέλετε να πουλήσετε τα κρασιά σας στην Ευρώπη, θα προσπαθήσουν οι Γάλλοι και οι Ιταλοί να το υπονομεύσουν, να το χύσουν στην ε, κυριολεξία, διότι είναι κακό το κρασί. Όχι, ίσα ίσα, επειδή είναι καλό το κρασί και είναι ανταγωνιστικό προς τα δικά τους το υπονομεύουν. Αλλά εντάξει, αυτό το είπε ένας παίκτη του χόκκι στον πάγο, έτσι, δεν είναι και καμιά αξιόπιστη πηγή. Εν πάση Θέλω να δώσω το λόγο στο Σερ Γκραμ Γότσον που είναι εισηγητής για τη Μολδαβία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τον Πρόεδρο. Είναι πολύ καλή ευκαιρία που έχουμε για να ενημερωθούμε για τα τεκτενόμενα στην Μολδαβία. Κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι πρόσφατα ε, λήφθησαν κάποιες αποφάσεις και την περασμένη εβδομάδα συμμετείχα και εγώ στην ψηφοφορία για τη θεώρηση διαβατηρίων και την απελευθέρωση στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ του Κοινοβουλίου και ελπίζω να πάει στην Ολομέλεια τώρα για να μπορέσουμε να εγκρίνουμε από κοινοβουλευτική σκοπιά το θέμα της απελευθέρωσης ε, θεωρήσεων διαβατηρίων. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, αν μου επιτρέπετε. Θα μπορούσατε να επεκταθείτε σε δύο-τρεις ε, τομείς που απλώς επιγραμματικά αναφέρατε στα σχόλιά σας. Είπατε και ενδιαφέρον το βρήκα ότι οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται αυτόν τον καιρό από την κυβέρνηση θα εγκαθιδρύσουν ε, μια κουλτούρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ελπίζω πάρα πολύ να γίνει αυτό, αλλά ε, θα μου επιτρέψετε να σας ρωτήσω αν η κυβέρνηση, εκτός από τις μεταρρυθμίσεις που διεξάγει αυτόν τον καιρό, μήπως προτίθεται επίσης να κάνει κάποιες μεταρρυθμίσεις ε, στο εκπαιδευτικό σύστημα στην παιδεία πώς χρησιμοποιείται η πολιτική του πολιτισμού και άλλοι τομείς που επηρεάζουν την κοινωνία για να ε, βοηθήσει να εγκαθιδεθεί αυτή η κουλτούρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τουλάχιστον ορισμένοι από εμά εδώ έχουμε ζήσει το εξή. Για να αλλάξει μια νοοτροπία, μια κουλτούρα χρειάζεται πολύ καιρό. Η δημόσια συμπεριφορά και η στάση του κόσμου υπολείπεται συχνά των επισήμων και νομοθετικών εξελίξεων σε μια χώρα. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε να προχωράει αυτή η διαδικασία και ποια πρόοδος έχει επιτευχθεί προς την κατεύθυνση αυτή. Επίσης, ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω λίγο περισσότερο για κάτι που επίσης θίξατε. Για μια θέση που έλαβε το Κοινοβούλιο πάρα πολύ σύντομα, που είναι το θέμα των σχολείων με λατινικούς χαρακτήρες στην υπερδνηστερία. Όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΑΣΕ και άλλοι προσπαθούν να αφήσουν αυτά τα σχολεία να εξακολουθήσουν να λειτουργούν χωρίς να ε, τους εμποδίζουν οι αρχές στην πρωτεύουσα της υπερνηστερίας ε, τη Ρασπόλ. Έχει υπάρξει καμία πρόοδο εκεί. Να μας πείτε και λίγο για τους γκαγκαούζους, γιατί πρόσφατα υπήρξαν κάποιες εξελίξεις κάπως ενοχλητικές και ανισχυτικές. Μήπως υπάρχει κάποια ξένη δύναμη που υποκινεί εκεί τα γεγονότα και θα μπορούσατε να μας πείτε τι γίνεται και με τους γκαγκαούζους. Αυτά περιορίζομαι, Πρόεδρε, γιατί υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να κάνουν και άλλες ερωτήσεις. Παρακαλώ. Thank uh, Σας ευχαριστώ και πάλι. Ο κύριος Κυρίλοφ, παρακαλώ. Πρόεδρε, διερωτάμε αν υπάρχει κάποιο από την Κομισιόν ε, να ακούσουμε πρώτα. Υπάρχει κάποιος εδώ από την Κομισιόν. Έχουμε κάποιον εδώ. No, <clears throat> Μάλιστα, ευχαριστώ. Νομίζω πως θα ήταν ε, καλό σε τέτοιες περιπτώσεις να έχουμε την γνώμη και την εικόνα από την Κομισιόν, της Κομισιόν μάλλον. Ε, καλωσορίζω την παρουσία του ομιλητή και πιστεύω πως είναι καλός ο σχεδιασμός να ακούσουμε και για την ε, Μολδαβία και για την Γεωργία. Έχω την εντύπωση πως μόλις τις αναταραχές στην Ουκρανία ξεχνάμε πως έχουμε σαφώς προτεραιότητες με τις δύο αυτές χώρες ώστε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσουμε και αν χάσουμε αυτήν την ε, προτεραιότητα θα ήταν πολύ, πολύ σοβαρό λάθος. Διότι έτσι θα δημιουργούσαμε πολλές αμφιβολίες, ε, προβληματισμό και θα ήταν πολύ κακό για την ε, πολιτική της Ένωσης. Πάντως, ούτως ή άλλως θα έπρεπε να το συζητήσουμε με την Κομισιόν και να προβούμε σε συγκεκριμένα και επίγοντα βήματα. Πώς να προγραμματίσουμε τα πράγματα, γιατί ε, βρίσκω πως ε, προχωράμε αργά. γιατι νομίζω πως ε, εξαρτάται από τον ταχύ ρυθμό η επιτυχία του εγχειρήματο αυτού. Νομίζω πως θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή στον εξυγχρονισμό και ένα πραγματικό πρόγραμμα δράσης. Είμαι βέβαιος ότι αυτό το σχέδιο, αυτή η δραστηριότητα θα έχει στήριξη από εδώ, από το Κοινοβούλιο. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να ακολουθήσουμε και γρήγορα βήματα από πλευράς κομισιών. Γιατί για την οικονομία Δεν έχουμε ακούσει κάποια καλή αξιολόγηση αρνητικών ε, ε, ε, εξελίξεων μετά από όλη αυτή τη διαδικασία που ξεκινήσαμε και θα πρέπει να το δούμε αυτό. Θα πρέπει να το δούμε αυτό πιο συνολικά, αντί να μιλάμε μόνο για εισαγωγές ίνου. Μάλιστα υπάρχει μεγάλη βουλγαρική κοινότητα στην ε, Μολδαβία που ασχολείται κυρίως με γεωργία και επεξεργασία των προϊόντων της, ε, φρούτα, λαχανικά αλλά και κρασί. Και φοβούνται ότι μάλλον θα χάσουν από αυτές τις νέες εξελίξεις. Απλά και μόνο λοιπόν για οικονομικούς λόγους πιστεύουν πως ε, ίσως η ε, Τελωνιακή Ένωση ήταν καλύτερη ιδέα. Δηλαδή προσπαθούμε να τα, να τα εξηγήσουμε αυτά, αλλά θα πρέπει ίσως ε, να ο κόσμος πια να δει τις προπτικές, τις εξελίξεις, να δει πού ε, προς τα πού κατευθύνονται για να δουν ε, ποια θα είναι η μοίρα τους. Πρέπει αυτό να το δούμε πιο ρεαλιστικά. Δεν είναι μόνο ένα καθεστώς άνευ θεωρήσεων, το οποίο και αυτό καλό είναι και πρέπει να προχωρήσει και αυτό σου γίνεται πιο γρήγορα, αλλά Εν γέννη θα ήθελα να υπάρξει μια συνέχεια σε αυτή την Επιτροπή και να κάνουμε μια πολύ καλή συζήτηση με τη συμμετοχή όλων των συναδέλφων, κρίσιμη μάλιστα συζήτηση όσον αφορά αυτές τις χώρες και τι θέλουμε να πετύχουμε για να δούμε τα αποτελέσματα πριν να λήξει η θητεία μας. Μέχρι τον Απρίλιο δηλαδή να ξέρουμε τι γίνεται με αυτές τις δύο χώρες, διότι θα υπάρξει αυτό το κενό μετά όπου δεν θα μπορέσουμε να ελέγξουμε και να παρακολουθήσουμε. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Kirillov. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κυρίλοφ. Η κυρία Ντάνοκα τώρα. Yes, thank you. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εδώ είμαι. Κύριε ε, ε, ε, πρόεδρε, εγώ είμαι αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις μας με τη Μολδαβία και θέλω να σας συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω για τις προσπάθειες που κάνετε και για τόσα μας είπατε. Παντού, σε όλους τους τομείς της δημόσιας και της πολιτικής ζωής. Η δική μου ερώτηση αφορά το εξής. Την καταπολέμηση της διαφθοράς στην οποία αναφερθήκατε. Ε, γι' αυτό έπεσε και η προηγούμενη κυβέρνηση άλλωστε. Έκτοτε τι ακολούθησε. Υπάρχει καμία προσπάθεια στην νομοθεσία για να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και διαπλοκή και μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου βίου. Τα γνωρίζουμε αυτά. Δυστυχώς αυτό έριξε την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν θέλω να επαναλάβω τις ερωτήσεις που έκαναν οι συνάδελφοί μου, αλλά με ενδιαφέρει και εμένα να μάθω και να ακούσω τη σκέψη σα για το δημοψήφισμα στην Καγκαουζία. Δεν αναφερθήκατε καθόλου σε αυτό. Επειδή είμαι και μέλος της Επιτροπής Ελευθεριών και σκιώδη συγγήτρια της ομάδας μου των Πρασίνων και της Ελεύθερης Ευρωπαϊκής Συμμαχίας, ε, μόνιμη συγγήτρια για ε, την ε, θεωρήσεις διαβατήριων και ιδιαίτερα τον κανονισμό 539 υποστηρίζουμε πλήρως ε, την μετάθεση της Μολαβίας στο παράρτημα 1 για άρση υποχρέωση θεωρήσεων διαβατήρια. Ξέρετε, το μεγάλο θέμα είναι τα βιομετρικά τώρα διαβατήρια. Η συγκήτρια ξέρετε ότι είναι η κυρία Τάνια Φαχιών πήγε στη Μολδαβία, από ό,τι ξέρω αυτό το Σαββατοκύριακο επρόκειτο να μεταβεί εκεί. Πώς προχωράει αυτή η διαδικασία αντικατάστασης των παλιών διαβατηρίων με βιομετρικά, ιδιαίτερα για τους κατοίκους της υπερδνηστερίας. Υπάρχουν προβλήματα να τους δοθούν διαβατήριο ή όχι. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κράισιλ παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε Κόρμαν, που είστε εδώ, γνωρίζετε πολύ καλά και το Μόναχο και τη Γερμανία ναι. και με καταλαβαίνετε. Μην αρχίσω τώρα τη διάλεκτο και σας προβληματίσω. Το 2008 ε, ζήσαμε την τεράστια τραπεζική και χρηματοπιστωτική κρίση που έπληξε όχι μόνο και σχεδόν ε, οδήγησε στην πτώχευση κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά δεν μας άφησε να έχουμε αρκετά χρήματα για να βοηθήσουμε καλύτερα και να επενδύσουμε περισσότερο ε, σε άλλες χώρες. Από παντού είναι το Ταμείο Μείων από όπου και να το πιάσει, ιδιαίτερα άμα δει κανεί τα οικονομικά και τα κοινωνικά προβλήματα σε ορισμένα κράτη-μέλη της ίδιας της Ένωσης. Ερωτώ λοιπόν, πόσο ισχυρά αυτό το κράχ ε, έπληξε τη χώρα σας. Τι μέτρα λάβατε για να το συγκρατήσετε κάπως ή να ανακουφίσετε αυτές ε, τις ε, συνέπειες. Έχω την αίσθηση ότι επίκειται το επόμενο κράχ τώρα άμα δει κανεί τις διεθνείς δραστηριότητες ορισμένων τραπεζών και άλλων οικονομικών παραγόντων. Ένα άλλο πολύ σημαντικό για την απελευθέρωση των διαβατηρίων είναι από μόνη τη σημαντική. Αλλά βλέπω στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιες τάσεις επανεθνικοποίησης και περιχαράκωση, και αρχίζω να ανησυχώ. Ορισμένοι θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτό το σύστημα, λένε. Αλλά οι εγκληματίες πάντα παρακάμπτουν τους κανόνες. Κάποιοι άλλοι που θέλουν να σπουδάσουν, να κάνουν ανταλλαγέ να εργαστούν, ακριβώς ε, φρενάρονται από αυτό το σύστημα. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε και στις ευρωεκλογές στις 25 Μαΐου εδώ στην Ένωση. Έχω μια ερώτηση για το εκπαιδευτικό σύστημα ακόμα. Γιατί στη Βαβαρία έχετε ζήσει καιρό και γνωρίζετε στη Γερμανία ότι υπάρχει αυτό το διτό σύστημα κατάρτισης. Ε, ξέρω ότι είναι διαφορετική επαγγελματική κατάρτιση στη χώρα σας, αλλά είναι σημαντικό για να μπορεί κανείς να είναι ανταγωνιστικό σε διεθνείς αγορές και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να προσελκύει επενδύσεις και στη βιομηχανία και στο εμπόριο χρειαζόνται πάντα ειδικευμένοι εργαζόμενοι άνδρες και γυναίκες στην ίδια τη χώρα που θέλω να επενδύσω. Ας πούμε, τι βήματα έχετε αναλάβει εκεί και ποια συνεργασία περιμένετε ή έχετε ήδη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το τομέα της παιδείας ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βουλιανίτς. Σας ευχαριστώ. κύριε Κόρμαν για τη σύντομη και ενδιαφέρουσα εισήγησή σας για την κατάσταση στη Μολδαβία. Εγώ είμαι σίγουρα υπέρ της διεύρυνσης. Νομίζω πως η πολιτική διεύρυνση είναι η πιο σημαντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η Ευρώπη δεν θα λειτουργήσει ως Ένωση μέχρι ότου να περιλαμβάνει όλες τις χώρες που θέλουν να ενταχθούν σε αυτήν και εσείς προφανώς και θέλετε να ενταχθείτε. Δεν υπάρχει, είπατε, δρόμος επιστροφής. Με χαρά το άκουσα αυτό. Άρα υπάρχει τρόπος να προχωρήσουμε και ελπίζω πραγματικά πως η Μολδαβία θα τα καταφέρει σε αυτή την πορεία. Εγώ θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήσεις. Υπάρχει προφανώς και είναι κατανοητό αυτό πίεση ε, ξανατολών. Ε, σαν αναφέρατε το θέμα των εξαγω... της εξαγωγής κρασιού, αλλά θα φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλοι τομείς ε, που ασκείται πίεση. Και θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας. Εσείς πώς τα βλέπετε, τι, πώς αισθάνεστε για όλα αυτά. ποια είναι η αίσθησή σας, ποια είναι η στάση του λαού σας απέναντι σε αυτή την πίεση. Η δεύτερη ερώτησή μου αφορά την ιδιωτικοποίηση. Εγώ συνήθως είμαι κατά της ιδιωτικοποίησης στις ε, χώρες ένταξης και για τους εξής βάσιμους λόγους. Μέχρι ότου να κατασταλάξει η χώρα ή ε, πολιτικά και κοινωνικά, η ιδιωτικοποίηση συνήθως καταλήγει σε φρικτές υποθέσεις διαφθοράς και άλλων ε, κακών. Στη χώρα σας ποια είναι η κατάσταση. Και πώς βλέπετε αυτή την παρότρινση για απόλυτη ιδιωτικοποίηση των πάντων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Κύριε ε, Ομιλητά, έχετε το λόγο, η σειρά σας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι για τις ενδιαφέρουσες αυτές ερωτήσεις. Δεν Ιδιαίτερα γιατί σταθερά υποστηρίζεται τη Μολδαβία στα διάφορα θέματα που συζητάτε εδώ. Θέσατε τρία ερωτήματα. Πρώτον, τη σημασία της παιδείας και του πολιτισμού. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί σας. Πρέπει να επενδύσουμε στην παιδεία και τον πολιτισμό. Βέβαια, τώρα περνάμε δύσκολη εποχή. Μια δύσκολη διαδικασία δηλαδή βελτιστοποίησης της παιδείας στη Μολδαβία τα τελευταία τρία χρόνια. Και δυστυχώς δεν μπορούμε πάντοτε να καταλήγουμε στη σωστότερη απόφαση και γι' αυτό μερικοί είναι δυσαρεστημένοι, παραμένουν δυσαρεστημένοι. Θα συνεχίσουμε όμως τις προσπάθειες γιατί η συζήτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ευρωπαϊκού μέλλοντος της Μολδαβίας δεν θα είναι δυνατή αν δεν προσέξουμε επαρκώς αυτό το σημαντικό τομέα. Τώρα στην υπερνηστερία. Δεν υπάρχει μόνο το θέμα των μολδαβικών σχολείων εκεί. Δυστυχώς βλέπουμε και άλλες προβοκάτσιες από την διοίκηση, την κυβέρνηση της υπερθενής Όπως η πρόσφατη σύλληψη ενός ε, διευθυντή κάποιου μολδαβικού σχολείου στην υπερδενιστερία και το λεγόμενο ultimatum που δόθηκε σε μία χείρα αστυνομικού στο Μπέλντερ. Υπάρχουν εμπόδια λοιπόν στη δημιουργία επικοδομητικού διαλόγου με τις αρχές του Τυρασπόλ. Το καλό είναι όμως ότι με το 5 συν 2 τα συζητάμε και ελπίζουμε αυτόν τον μήνα να ξαναγίνει συνάντηση. Είναι καλή μέθοδος αυτή για τη συζήτηση των τρεχόντων προβλημάτων. Το κακό είναι ότι δεν έχει επισυμβεί καμία πρόοδος στις διαπραγματεύσεις αυτές. Δεν θέλουν να συζητήσουμε το θέμα της πολιτικής λύσης της διαμάχης αυτής. Μόνο τεχνικά προβλήματα όπως τα σχολεία στην υπερνηστερία. Νομίζω όμως ότι, ότι σωστή είναι η συμπεριφορά των μολδαβικών αρχών να επιδεικνύουν πνεύμα επικοδομητικό και όχι αρνητικό και να προσπαθούν να ακόμη και απλώς να διατηρήσουν υποέλεγχο την κατάσταση και εκτιμούμε ιδιαίτερα την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων εταίρων στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Για την καγκαουζία Πράγματι δεν την ανέφερα στην παρουσίασή μου. Αλλά με τα χαράς να σας πω τι συμβαίνει σε αυτή την περιφέρεια της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Υπάρχουν προβλήματα που προέρχονται από το παρελθόν. Οι αρχές του Κομράτ που είναι η πρωτεύουσα της Γαγαουζίας έχουν παράπονα για τη σχέση με τις κεντρικές αρχές. Επίσης, για την μολδαβική νομοθεσία και το ειδικό καθεστώς της Γαγαουζίας. Και οι κομμουνιστές επίσης ήταν στην εξουσία 8 χρόνια και δεν κατάφεραν δεν πρόσεξαν αρκετά την κατάσταση εκεί της αυτόνομης αυτής περιοχής και τώρα, τώρα η κατάσταση προκύπτει διότι έχουμε βουλευτικές εκλογές τον Νοέμβριο και εκείνοι επίσης στη Γαγαουζία σε ένα χρόνο θα πρέπει να ελέγξουν τον Μπασκάν, τον πρωθυπουργό τους. Και ορισμένα κόμματα, κεντρικά κόμματα, θέλουν να παίξουν παιχνίδια σε αυτό το θέμα. Τώρα γίνεται λόγος για το λεγόμενο δημοψήφισμα που έγινε στην Γαγαουζία πριν από δύο εβδομάδες. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν παράνομο διότι δεν συμφωνούσε με τον νόμο ούτε με τις προβλέψεις της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής της Μολδαβίας αλλά αποφασίσαμε να μην προκαλέσουμε πρόβλημα και να ζητήσουμε από τους Γαγαούζους επικοδομητικό διάλογο Έγινε και μια επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Γαγαουζία, συζήτησε με όλες τις τοπικές αρχές και αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μια ειδική επιτροπή του Κοινοβουλίου για να αρχίσει διάλογος ως προς τα νομοθετικά και νομικά προβλήματα και θα δημιουργηθεί και μια ομάδα εργασίας για ένα αναπτυξιακό σχέδιο της αυτόνομης περιοχής τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Νομίζουμε ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος βήμα-βήμα να συνεννοηθούμε μαζί τους και ελπίζουμε ότι αυτή η προσέγγιση των κεντρικών αρχών θα γίνει δεκτή και από τους αυτόνομους. Τώρα κύριε Κυρίλοφ μου, Μιλήσατε για την κατάσταση στην Ουκρανία. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι η Ουκρανία είναι πολύ σημαντική χώρα για μας. Είναι γείτονά μας και πολύ σημαντικός οικονομικός εμπορικός εταίρος μας και ανησυχούμε για τις εξελίξεις εκεί. Ελπίζουμε ότι οι προσπάθειες και της Ένωσης και άλλων παραγόντων θα καταλήξουν σε μια σταθεροποίηση. Ελπίζουμε δε η Ουκρανία να συνεχίσει δημοκρατικά να εξελίσσεται και να έχει δικαίωμα να αποφασίσει για το μέλλον του ο λαός. Εμείς δεσμευόμαστε γι' αυτό, τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα υποστηρίζονται από μας και θα συνεχίσουμε αυτόν τον ρόλο να παίζουμε. Βεβαίως έχετε δίκιο κύριε Κυρίλοφ. Το θέμα δεν είναι μόνο το κράσι. Το κρασί είναι απλώς ένα παράδειγμα του πόσο γρήγορα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρθηκε. Έχετε δικαίωμα όμως, έχετε δίκιο, προετοιμάζουμε τώρα τη συμφωνία για τον χώρο ελεύθερων συναλλαγών και αφού εγκριθεί το πρόγραμμα σύνδεσης θα διαμορφώσουμε ένα εθνικό σχέδιο τις επόμενες εβδομάδες και μήνες και εκτιμούμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι υπάρχει δυνατότητα να μπούμε και στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης πράγμα που θα μας επέτρεπε τους παραγωγούς μας στη Μολδαβία να έχουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκά ταμεία για να προετοιμαστούν και να είναι πιο ανταγωνιστικοί. Η Συμφωνία Σύνδεσης και Ελεύθερων Συναλλαγών ευνοεί την Μολδαβία διότι πρόκειται για ασυμμετρική συμφωνία και άρα για ευαίσθητους τομείς έχουμε 7, 8, 9 χρόνια καιρό να προετοιμαστούμε ώστε οι παραγωγοί μας να μπορέσουν να ανταγωνιστούν τους ενωσιακούς. Προς στιγμή 50% των αγαθών μας εξάγονται στην Ένωση και είμαστε βέβαιοι ότι η Συμφωνία Σύνδεσης θα μας επιτρέψει να αυξήσουμε τις εξαγωγές μας στην Ευρωπαϊκή Αγορά. Ελπίζουμε να ε, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε μάλλον να υπάρξουν και καινούργια προβλήματα και αδυναμίες αλλά αν η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιδράσει το ίδιο γρήγορα όπως το έκανε με το κρασί νομίζω ότι θα τα βγάλουμε πέρα. Κυρία Σδανόκα, μίλησε για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Είναι πολύ σημαντικό θέμα στη Μολδαβία η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και η καταπολέμηση της διαφθοράς. Πέρυσι το Δεκέμβριο στη Βουλή εγκρίναμε μια δέσμη μέτρων ακριβώς για το θέμα αυτό της δικαστικής μεταρρύθμισης και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Υπάρχει το θέμα ας πούμε της ε, επαγγελματικής ακαιρεότητας των δικαστών από τη μία, από την άλλη όμως αποφασίσαμε να αυξήσουμε και τους μισθούς τους. Δεν είναι πολύ καλή απόφαση για τους πολίτες μας γιατί δεν καταλαβαίνουν γιατί να αρχίσουμε από αυξήσεις μισθών δικαστών αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος μετά από διαβουλεύσεις και με διεθνείς εμπειρογνώμονες αποφασίσαμε να πάρουμε αυτό το μέτρο και θα δούμε τώρα πώς μπορεί να εφαρμοστεί. Θα προσέξουμε ιδιαίτερα και αρχίσαμε επίσης ε, μια ομάδα εργασίας στη Βουλή μας μας υποστήριξε και η Επιτροπή Βενετίας και τους επόμενους μήνες θα εγκριθούν και, άλλοι, και άλλα νομοσχέδια ε, ε, για την εισαγγελία και τις ιδιοκτικές αρχές. Ε, θα δημιουργήσουμε επίσης ένα κέντρο καταπολέμησης της διαφθοράς και μια Εθνική Επιτροπή για την Ακαιρεότητα η οποία θα ασχοληθεί θα αποτελείται μάλλον από υψηλόβαθμους αξιωματούχους ε, και βουλευτές και ελπίζουμε να αρχίσουμε τη μεταρρύθμιση όχι από τους πολίτες αλλά από το ανώτερο επίπεδο. Τα βιομετρικά Ειδικά διαβατήρια τώρα και η απελευθέρωση των θεωρήσεων. Σας βεβαιώνω ότι είμαστε προετοιμασμένοι 100%. Και οι αρχές μας είναι ικανές να διασφαλίσουν την χορήγηση βιομετρικών διαβατηρίων για όλους τους πολίτες. Πολλοί τα έχουν ήδη. Και νομίζω ότι ήδη πάνω από 15.000 το μήνα θα εκδίδονται. Τα ίδια και για τους πολίτες της υπερθυνιστερίας. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του θέματος ε, του, από την Ευρώπη που ήρθε στη Μολδαβία επίσης διαπίστωσε ότι υπάρχει πρόοδος σε αυτό. Κύριε Κρέσεντορφερ, στα γερμανικά με ρωτήσατε για την χρηματοοικονομική κρίση το 2008 και πώς έπληξε τη Μολδαβία και πώς έχουν οι εξελίξεις αυτές το τελευταίο διάστημα. Γνωρίζετε κύριε Κράσελντορφερ ότι τότε δεν μας ε, έπληξε το πρώτο κύμα ήδη αυτό το 2008 διότι η Μολδαβία δεν είχε εκεί καμιά τρομερή οικονομική δραστηριότητα σε αυτά τα θέματα της κτήματα αγοράς και οικοδομών. Αλλά το δεύτερο κύμα μας έπληξε σφοδρότατα το 2009. Είχαμε και βουλευτικές εκλογές δύο φορές εκείνο το χρόνο και το μεγαλύτερο επίτευγμα της κυβέρνησής μας είναι ότι τότε καταφέραμε το 2010 κάπως να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση. Βεβαίως εργαζόμαστε πολύ στενά ε, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεργασία προβλήματα υπάρχουν, δεν το αρνούμε το τελευταίο διάστημα και είναι επίκαιρο το θέμα και τώρα στο Κοινοβούλιο, διότι προετοιμαζόμαστε να κάνουμε όλα τα απαραίτητα βήματα στο Κοινοβούλιο, στην νομοθεσία όλες τις αλλαγές, για να ε, σταθεροποιήσουμε το χρηματοοικονομικό καθώς και τον πιστοτικό και τον τραπεζικό τομέα. Το πλεονέκτημά μας είναι ότι παραμένουμε σε στενή επαφή με το Δούνου του και άλλους ε, διεθνείς ε, οικονομικούς οργανισμούς που μας παρέχουν πραγματογνωμοσύνη και υποστήριξη. Επίσης αναφέρατε το θέμα της απελευθέρωσης των διαβατηρίων, ε, το θεωρήσεων δηλαδή και ότι ανησυχούν οι ευρωπαϊκές χώρες για τις εργασίες. Κοιτάξτε, αυτοί, όλοι οι Μολδαβοί δηλαδή που θέλουν να φύγουν από τη χώρα την έχουν ήδη καταλήψει. Και βέβαια γνωρίζουν οι πολίτες μας ότι η απελευθέρωση των θεωρήσεων πλέον μας επιτρέπει να κινούμεθα ελεύθερα. Μόνο να ταξιδεύουμε, όχι να εργαζόμαστε παντού στην Ένωση. Το ξέρουν οι πολίτες, τους ενημερώνουμε πάρα πολύ. Είναι περισσότερο ψυχολογικό το επιχείρημα. Και βεβαίως στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τις ε, προϋποθέσεις εκείνες για εργασία για τους πολίτες μας στην ίδια μας τη χώρα. Να μην φεύγουν οι Μολδαβοί. Και ε, το επόμενο ερώτημά σας ε, για τους επενδυτές το τελευταίο διάστημα έχουμε πολύ σοβαρούς επενδυτές και βαβαρούς και γερμανούς. Drexel Mayer για παράδειγμα είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται πάρα πολύ. Έχουμε και δημιουργήσει ειδική ελεύθερη ζώνη για την εταιρεία αυτή και έρχονται και άλλοι επενδυτέ από τη Γερμανία. Προσεχώς και η Λεόνη που είναι άλλη μεγάλη σημαντική εταιρεία. Δημιουργούνται και χιλιάδες θέσεων εργασίας έτσι. Ελπίζουμε πάρα πολύ Συμφωνία Σύνδεσης και η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών να βοηθήσει για να δώσει το πράσινο φως και για άλλους επενδυτές. Ε, κατανοούμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό είναι ο σωστός δρόμος. Καλή νομοθεσία, καλό επιχειρηματικό κλίμα στη χώρα, περισσότερες επενδύσεις και τότε θα μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτή την εξέλιξη που μεταναστεύει ο κόσμος. Και ελπίζω πάρα πολύ να επαναπατηθούν οι Μολδαβοί που βρίσκονται εκτός της χώρας αυτόν τον καιρό. Εκεί συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τη λεγόμενη εταιρική σχέση για την κινητικότητα. Και λειτουργεί αυτό βήμα-βήμα με καλά αποτελέσματα ήδη. Δύο ακόμα τελευταία ερωτήματα για τη σχέση μας με τη Ρωσία. Στα αγγλικά. Ρωτήσατε ε, για τη σχέση μας με τη Ρωσία. Ε, θα ήθελα να πω το εξής. Βεβαίως η Ρωσία είναι πάρα πολύ σημαντικός εταίρος για μας. Το 20% των εξαγωγών μας πηγαίνουν στη ρωσική αγορά. Εισάγουμε 100% φυσικό αέριο από τη Ρωσία. 100.000 εργαζομένους έχουμε στη Ρωσική μοσπονδιά Μολδαβούς εργάτες. Και βεβαίως η Ρωσία είναι σημαντικός ε, παράγων όταν ε, πρέπει να συζητήσουμε το θέμα της ε, πολιτικής διένεξης της υπερθυνιστερίας. Όπως σας είπα και προηγουμένως, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να διατηρήσουμε το διάλογο με τη Ρωσία, τη Μόσχα. Και πιστεύουμε ότι η απόφαση που λάβαμε να αναπτύξουμε τη χώρα μας κατά το ευρωπαϊκό μοντέλο δεν θα πρέπει να αποτελεί αντίφαση ε, για τη συνεργασία μας με όλους τους ε, ξανατολών εταίρους ε, της Ρωσίας συμπεριλαμβανομένης. Όταν το συζητούμε μαζί τους δεν διαφωνούν και προσωπικά είχα συζητήσεις με τους συναδέλφους από την κρατική δούμα, τη Ρωσική Βουλή. Πώς μπορεί να διαφωνήσει κανείς ότι είναι κυρίαρχη απόφαση της Μολδαβίας κάτι τέτοιο. Από την άλλη, βέβαια, δεν μπορούμε και να είμαστε απροετοίμαστοι για ενδεχόμενα αρνητικά γεγονότα και εξελίξεις φέτος. Και το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν μπορούμε να εξαγάγουμε τα κρασιά μας. Πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια χάσαμε πέρυσι. Ελπίζω να μην ξανάχουμε έχουμε τέτοιες εκπλήξεις το 2014 σε ό,τι αφορά τα νοπάω οποροκυπευτικά μας. 80% τα εξάγουμε στη ρωσική αγορά. Θα συνεχίσουμε λοιπόν το διάλογό μας. Βεβαίως υπάρχουν πάντα θέματα γεωπολιτικών ανταγωνισμών στην περιφέρεια και το κατανοούμε, αλλά προσπαθούμε να έχουμε έτσι, μια επικοδομητική στάση και συμπεριφορά και φέτος. Και όπως σας είπα, ακόμα και αν έχουμε κάποια προβλήματα ελπίζουμε να μπορέσουμε να τα ξεπεράσουμε και να προσβλέπουμε και στη δική σας υποστήριξη και συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι έχει η κατάσταση. Επίσης, ρωτήσατε για τη διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων στη Μολδαβία. Να σας ενημερώσω πάρα πολύ σύντομα σχετικά. έχουμε πάνω από 90% ιδιωτικοποίηση. Υπάρχουν ακόμα και μεγάλες όμως κρατικές εταιρείες. Τώρα είναι και προεκλογική χρονιά, μάλλον ένας χρόνος πριν τις εκλογές και το περιβάλλον δεν είναι πάρα πολύ θετικό ούτε γενικά η κατάσταση στην περιοχή μας. Δεν έχουμε πάρει οριστικές αποφάσεις ε, ως προς το θέμα του αν θα πρέπει να συνεχιστούν οι ιδιωτικοποίησει, Αλλά πάνω από 90% επαναλαμβάνω έχουν ήδη αποκρατικοποιηθεί εταιρείε και είμαστε σε καλό δρόμο νομίζω όταν συζητούμε για θέματα ελεύθερης αγοράς κτλ. Okay, thank you very much, Mr. Speaker. Um, our colleagues... Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως είδατε, Πολλές ερωτήσεις υποβλήθηκαν και όλες αναφέρονταν σε συγκεκριμένα προβλήματα. Ε, σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι εξακολουθούμε να στηρίζουμε τις προσπάθειες της χώρας σας από το Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε πολύ. Again, I would like to thank you. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας. Θα ήθελα να ε, ευχηθώ ε, καλή επιτυχία σε όλους για τις ευρωεκλογές και ελπίζω ότι μετά από τον Νοέμβριο θα ξανασυναντηθούμε για την μια φιλοευρωπαϊκή ε, κυβέρνηση στην Μολδαβία και το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. σε <clears throat> Uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε την ε, σημερινή απογευματινή μας συνεδρίαση και με χαρά καλωσορίζω την ε, εξοχότητά της, κυρία Μάγια Πανζικίτσε, που είναι υπουργό Εξωτερικών της Γεωργίας, μιας χώρας που είναι προσιλωμένη στην ευρωατλαντική ολοκλήρωση και που είναι στην πορεία για επίτευξη αυτών των στόχων. Ε, θα σας δώσω λοιπόν το λόγο για να μας κάνετε μια εισήγηση για 10-15 λεπτά και σίγουρα οι συνάδελφοι θα σας υποβάλουν ερωτήσεις στη συνέχεια. Έχετε το λόγο λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι. Είμαι εξαιρετικά ευτυχή ε, και αισθάνομαι μεγάλη τιμή που μπορώ σήμερα να μιλήσω ενώπιον τη ε, επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου. Σα ευχαριστώ για αυτή τη μοναδική ευκαιρία να σα μιλήσω σήμερα εδώ για τι προπτικές και προκλήσει τη Ευρωπαϊκής, ε, της Γεωργίας στην πορεία προ την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Θα ήθελα επίση να σα ευχαριστήσω για τη ισχυρή στήριξη του Ευρωκοινοβουλίου προ τη Γεωργία και στα, μέσω των πολυάριθμων ψηφισμάτων σα. Η αφοσίωσή σα και καθενός χωριστά αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο συνολικά οδηγεί στην καρποφόρα και επιτυχή μας συνεργασία. Σας διαβεβαιώ πως οι συστάσεις σας και οι συμβουλές σας είναι μεγάλη σημασία για τη χώρα μου που προσπαθεί να δημιουργήσει μια γνήσια ευρωπαϊκή δημοκρατία και να αποκαταστήσει τη θέση της στην κοινή ευρωπαϊκή οικογένεια. Η συνθήκη της Λισαβόνας για την Ευρωπαϊκή Ένωση προώθησε σημαντικές αλλαγές στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένου κυρίως για το Ευρωκοινοβούλιο, ε, το οποίο η φωνή είναι πιο ισχυρή μέσω αυξημένων αρμοδιοτήτων και αυξημένου ρόλου στο σύνολο του ευρωπαϊκού ε, ε, αρχιτεκτονήματος. Έχοντας όλα αυτά υπόψη, ε, αγαπητοί μου φίλοι, θα βασιστούμε στην περαιτέρω στήριξή σας για, την Ευρω... για τη Γεωργία και τις ευρωπαϊκές της ε, βλέψεις. Καλωσορίζουμε κάθε δυνατότητα για ανοιχτό διάλογο μαζί σας για όλα τα θέματα των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωργίας. Και τώρα επιτρέψατε μου να συνεχίσω μοιραζόμενοι μαζί σας ε, το agenda Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Γεωργιανής Κυβέρνησης με βάση σημαντικές και ξένες εξελίξεις ε, στην ε, χώρα μου. Ε, θα μιλήσω και για εξωτερικούς παράγοντες και τέλος θα σας παρουσιάσω τις προσδοκίες της Γεωργίας όσον αφορά τη διάσκεψη κορυφής της Ρήγας το 2015 μέσα στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Η ευρωπαϊκή και η ευρωατλαντική ολοκλήρωση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της εξωτερικής πολιτικής αλλά και της εγχώριας πολιτικής της Γεωργίας. Είναι ένα εθνικό ιδεώδες το οποίο στηρίζει ο γεωργιανός λαός και όλα τα βασικά πολιτικά κόμματα. Το αποτέλεσμα των ε, προεδρικών εκλογών του Οκτωβρίου 2013 απέδειξαν ε, περίτρανα τις ευρωπαϊκές προσδοκίες του λαού της Γεωργίας. Ταυτόχρονα ε, γνωρίζουμε απόλυτα πως η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι μια συνεχιζόμενη εσωτερική διαδικασία όπου εμπλέκονται ε, αλλαγές και μεταρρυθμίσεις μεγάλης κλίμακας. Από την ανάληψη του, της εξουσίας του, τον Οκτώβριο του 2012 η κυβέρνησή μας ξεκίνησε και εφάρμοσε βασικές πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις που στόχο έχουν την ενίσχυση της δημοκρατίας, το κράτο δικαίου, την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος, ανθρώπινα δικαιώματα και ε, ελευθερίες, στήριξη των επιχειρήσεων και της κοινωνικής πρόνοιας. Το 2013 ήταν ένα έτος γεμάτο από διάφορα ξεμνημόνευτα γεγονότα και επιτεύγματα της Γεωργίας. Για να συντομεύσω θα τονίσω μόνο ε, κάποιες κάποια βασικά επιτεύγματα στην εσωτερική μας πολιτική. Καταρχήν η Γεωργιανή Δημοκρατία προχωρά στο επόμενο βήμα της δημοκρατικής εξηγίασης. Οι, οι εκλογές του Οκτωβρίου παρακολουθήθηκαν από ε, διεθνείς οργανισμούς και θεωρήθηκαν ελεύθερες και δίκαιε. Επίση, ο γεωργιανός λαός ε, σε κατέστησε σαφέ ότι δεν θα δεχθεί πλέον αποκλήσεις από το δημοκρατικό μονοπάτι της ανάπτυξης και νομίζω πως αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά μας επιτεύγματα. Ακόμα ένα ορόσημο για την εξυγίανση τη δημοκρατική είναι οι πρόσφατες συνταγματικές μεταρρυθμίσεις που δημιούργησαν ένα σύγχρονο σύστημα ισορροπιών ανάμεσα στο εκτελεστικό και στο ε, πολιτικό κομμάτι της εξουσίας, ε, ώστε να ενισχυθεί η αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Επίσης κατεβλήθησαν προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η απόλυτη ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος. Τα δικαστήρια αποκτούν και πάλι την εμπιστοσύνη και το σεβασμό του λαού. Αυτή τη στιγμή τα γεωργιανά μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ελεύθερα από πολιτικές πιέσεις όπως και στις υπόλοιπες δημοκρατίες. Η προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων είναι ανάμεσα στις βασικές μας προτεραιότητες. η Εθνική Στρατηγική Περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύθηκε πρόσφατα και παρουσιάστηκε και θα υιοθετηθεί από την κυβέρνηση αυτή την εβδομάδα. Σε αυτό το πλαίσιο είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονε για την πολύτιμη συμβολή του Συμβούλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ε, μειονότητες του Τόμας Χάνεμπεργκ. Τέλος, η Γεωργία είναι μια χώρα όπου το επιχειρήν είναι εύκολο και όπου οι επιχειρήσεις λειτουργούν ελεύθερα σε ένα ανταγωνιστικό ε, περιβάλλον με ισχυρές εγγύησεις για τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Παρά τις οικονομικές προκλήσεις, η στήριξη για την κοινωνική πρόνοια έχει διπλασιαστεί, ε, έχει εισευθεί ασφάλεια για όλους και νέος κώδικας εργασίας σύμφωνα έχει επίσης επικυρωθεί σύμφωνα με τα στάνταρ του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Στόχο έχουμε να εξασφαλίσουμε μακροπνοή ε, οικονομική ανάπτυξη για τη γεωργία για όλους. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Διεθνούς Τράπεζας, ε, η γεωργία αναπτύσσεται κατά 5 ή 6% μέσα στο 2014. Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών της κυβέρνησης και των σταθερών ευρωπαϊκών βλέψεων του γεωργιανού λαού, το 2013 ήταν εξαιρετικά επιτυχές για τις σχέσεις μεταξύ Ένωσης και Γεωργίας. Καταρχήν, στη διάσκεψη κορυφής του Βίλνιους για την Ανατολική Εταιρική Σχέση, ξεκινήσαμε συμφωνία συνεργασίας, σύνδεσης συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματο μιας περιοχής ελευθέρων συναλλαγών. Αυτό το θεωρούμε ως ένα βασικό πρόγραμμα για την οργάνωση της χώρας μας και αντιπροσωπεύει μια βασική μετακίνηση όσον αφορά τις πολιτικές προοπτικές αλλά και τις οικονομικές προοπτικές καθώς και την οικονομική ολοκλήρωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυξάνεται η αποτελεσματικότητα της γεωργίας ως ε, προορισμός επενδύσεων επενδύσεων, ανοίγοντας μεγαλύτερες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις. Αναμένω πως αυτές οι νέες πραγματικότητες θα ε, γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευση από την Γεωργιανή αλλά και τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα. Ακόμα ένα μέγα επίτευγμα τη διάσκεψη κορυφή του Βίλνιου ήταν η υπογραφή του πλαισίου για τη συμμετοχή τη Γεωργία σε επιχειρήσει, σε διαχείριση τη κρίση τη Ένωση, πράγμα το οποίο φέρει βασικά ένα πολύ ισχυρό μήνυμα Δηλαδή, η συμμετοχή μας σε πολιτικές και στρατιωτικές αποστολές και οι δέσμευσή μας αυτές ε, σημαίνει πως η Γεωργία δεν χαίρει μόνο των ε, ρυθμίσεων της Ένωσης για την ασφάλεια, αλλά θεωρείται και ως αξιόπιστος εταίρος της προσπάθειας της Ένωσης να οικοδομήσει ειρήνη και ασφάλεια παγκοσμίως. Έχουμε σημειώσει δε σημαντική πρόοδο προς την ολοκλήρωση της πρώτης νομοθετικής φάσης ε, όσον αφορά το πρόγραμμα δράση για την απελευθέρωση των θεωρήσεων, το οποίο θεωρήθηκε θετικά από την ε, Κομισιόν, αυξημένη κινητικότητα, η εισαγωγή ενός ελεύθερου θεωρήσεων καθεστώτος θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας για τους απλούς πολίτες της Γεωργίας. Γι' αυτό η κυβέρνησή μου είναι αποφασισμένη να μην φυστεί προσπαθειών ώστε να επιτύχει αυτό το στόχο μέχρι την διάσκεψη κορυφής της Ρήγας για την ανατολική εταιρική σχέση. Εν τω μεταξύ θα πρέπει να σκεφτούμε όμως και τις προκλήσεις που συνοδεύουν αυτήν την διαδικασία. Πρώτη προτεραιότητα για τη Γεωργία είναι να υπογράψει την Συμφωνία Σύνδεσης Ένωσης Γεωργίας όσο γίνεται πιο σύντομα. Καλωσορίζουμε την ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσει την υπογραφή της συμφωνίας αυτής πριν το φθινόπορο. Από την πλευρά μας κάνουμε ό,τι χρειάζεται ώστε αυτό να υλοποιηθεί. Το δεύτερο σημείο που θέλω εδώ να παρατηρήσω είναι ότι είμαστε περισσότερο από ποτέ αποφασισμένοι να μεταφράσουμε αυτήν τη δέσμευση σε συγκεκριμένες ενέργειες και πολιτικές προς όφελος των πολιτών μας. Ε, είμαστε αποφασισμένοι να αντιδικοποιήσουμε τις προσπάθειες μεταρρύθμισης ώστε να προετοιμαστεί ένα στέρεο έδαφο για την εφαρμογή της συμφωνία σύνδεση, που είναι πιο περίπλοκη και απαιτητική διαδικασία. Επιτά οι νέε πραγματικότητε που θα υπάρξουν, ισχύσουν μετά από την υπογραφή της Συμφωνίας σύνδεση. Επίση σημαίνουν ε, συνολικέ και δαπανηρέ μεταρρυθμίσει που έχουμε αναλάβει να υλοποιήσουμε. Προς αυτό το σκοπό η κυβέρνησή μας άρχισε να σχεδιάζει μια, προ... μια ατζέντα μεταρρυθμίσεων υπό το φως των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συμφωνία Σύνδεσης. Είμαστε έτοιμοι να εγκαίρως να υλοποιήσουμε την ατζέντα για την ε, σύνδεση. Πιστεύουμε πως οι προσπάθειές μας θα στηριχθούν ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τις αρχές more for more. Περισσότερα για περισσότερα. Σε αυτή τη γραμμή θα ήθελα να καλωσορίσω την πρόσφατη δήλωση του Επιτρόπου Φίλε στην διάσκεψη για την ασφάλεια στο Μόναχο. Η προοπτική ε, ένταξη στην Ένωση είναι ένα φως στο τέλος του τούνελ, όπως το έθεσε και ο Επίτροπος, και αυτός είναι ένα καταλήτης για τις μεταρρυθμίσεις ε, για τις χώρες δηλαδή της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, περιλαμβανομένης και τη Γεωργία. Η δέσμευσή μα είναι να δείξουμε απτή πρόοδο στην πορεία του εξυγχρονισμού και του εξευρωπαϊσμού της Γεωργία και ελπίζουμε πω η Ένωση τελικά θα δείξει την αποφασιστικότητά της και θα αναγνωρίσει το ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας μου καθώς και αυτό των άλλων ε, ε, των άλλων ε, χωρών της Ανατολικής ε, ε, εταιρικής σχέσης. Ε, χρειάζεται αλληλεγγύη και στήριξη όσο γίνεται περισσότερο σε σχέση με τους εξωτερικούς παράγοντες. Διάφοροι ε, εταίρια ε, της Ανατολικής Ευρώπης περιλαμβανομένες της Γεωργίας δέχονται αυξανόμενη πίεση από τη Ρωσική Ομοσπονδία, ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, ώστε να αναθεωρήσουν τις ευρωπαϊκές τους βλέψεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν μεταξύ των πρώτων που στάθηκε όρθος στο ανάστημά του και καταδίκασε τις ρωσικές ενέργειες στο ψήφισμα του του Σεπτεμβρίου 2013 και χρησιμοποίησε κάθε ευκαιρία για να επαναλάβει τις ανησυχίες του για αυτό το θέμα μέσα στο πλαίσιο άλλων ψηφισμάτων. Δεν τρέφουμε αυταπάτες όσον αφορά τη δυνατότητα περαιτέρω προκλητικών ενεργειών της Μόσχας, ιδιαίτερα πριν από την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης. Ωστόσο, με συγχωρείτε. Ωστόσο θα επαγρυπνούμε ώστε να εμποδίσουμε οποιαδήποτε κλιμάκωση που μπορεί να εμποδίσει την συνυπογραφή, την εφαρμογή της συμφωνίας. Είμαστε έτοιμοι να σταθούμε, <laughs> αντισταθούμε σε κάθε πίεση, διότι τα όσα διακυβεύονται δεν είναι ακόμα μια διεθνή συμφωνία, αλλά το ευρωπαϊκό μέλλον της Γεωργίας. Ταυτόχρονα θα πρέπει να αποκομίσουμε διδάγματα από τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλο της το κύρος, το βάρος, ώστε να εμποδίσει επεμβάσεις από τρίτα μέρη στις σχέσεις της με τους ε, εταίρους της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Θα πρέπει να σχεδιάσουμε μια κοινή θέση ώστε να ασκήσουμε ώστε μάλλον να αντισταθούμε στα καταναγκαστικά μέτρα που λαμβάνονται έναντι των εταίρων της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Θα πρέπει να στηρίξουμε τη βασική αρχή της μη παρέμβασης και των ε, κυρίαρχων δικαιωμάτων κάθε, της κάθε χώρας να ασκήσει την ε, ε, εξωτερική της πολιτική. Κυρίες και κύριοι, τα τελευταία χρόνια η Γεωργία προσπαθεί να περιορίσει τις εντάσεις με την ε, Ρωσία και ήμασταν συνεπείς στις προσπάθειές μας. Η προηγούμενη κυβέρνηση ανέλαβε να μην χρησιμοποιήσει βία ε, κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Γεωργία εισήγαγε το ε, καθεστώς ε, άνευ θεωρήσεων για τους πολίτες της Ρωσίας και στήριξε την ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ. Για να περιοριστούν οι εντάσεις αρχίσαμε να διερευνούμε τους διάφορους τομείς συνεργασίας που να μην επιβαρύνουν όμως την κυριαρχία και την διαθεκία κυριότητα της Γεωργίας. Πετύχαμε κάποια αποτελέσματα όπως ας πούμε το άνοιγμα ε, το σταδιακό των ρωσικών αγαρών για τα δικά μας προϊόντα και οι σχέσεις μας έχουν εντατικοποιηθεί. Λάβαμε και δε την απόφαση να συμμετέχουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σότσι. Η προσέγγιση μας ήταν σαφές, σαφής όταν λάβαμε αυτή την απόφαση ότι δηλαδή θα πρέπει να αναμεγνύεται ο αθλητισμός με την πολιτική. Ωστόσο, σε απάντηση σε αυτά τα βήματα, η Ρωσική Ομοσπονδία αντίθετα προσπάθησε να κατευθύνει και να χρησιμοποιήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σότσι κατά της εδαφικής ακυριότητας της Γεωργίας, κυρίως προωθώντας το υποτιθέμενο καθεστώς αυτονομίας των κατεχόμενων περιοχών της Γεωργίας, καθώς και τη δημιουργία ε, μιας ε, ζώνης ε, ασφάλειας στην περιοχή της γεωργίας που βρίσκεται, στον Κάφκασο, μια ελεγχόμενη ζώνης σε μήκους 11 χιλιόμετρων. δεν μας επηρέασαν όμως όλα αυτά και παραβαίνοντας τη διεθνή νομοθεσία καθώς και το πάυση του πυρός η Μόσχα συνεχίζει τις καταστροφικές της δραστηριότητες, σε σειρματοπλέγματα στη γραμμή ε, κατοχής. Καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή για τους τοπικούς πληθυσμούς. Περιμένουμε δε και άλλες ενέργειες από την πλευρά της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αυτή η παράνομη διαδικασία, αφού έπαψε λίγο λόγω της ε, διεθνούς κατακραυγής, ξανασυνεχίζεται τώρα και παραβιάζοντας τα θεμελιώδη δικαιώματα των τοπικών πληθυσμών μέσω τεχνητών ε, ε, συνόρων έχει ήδη διεισδύσει 15 χιλιόμετρα και έχει προκαλέσει ανθρωπιστικά προβλήματα για πολλές οικογένειες. Περιμένουμε δε περαιτέρω προσπάθειες των Ρώσων για να αυξήσουν τις πιέσεις στην Γεωργία. Η κυβέρνησή μας συνεχίζει να συνεργάζεται στενά με την Ένωση και άλλους διεθνείς εταίρους αλλά και φιλικά έθνη ώστε να αποφύγει και να αποτρέψει περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης η πολιτική στήριξη αλλά και οι δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα ψηφίσματά του που καταδικάζουν τις αναφερόμενες, προαναφερθήσεις μάλλον παράνομες διαδικασίες είναι πολύ σημαντικές. Το 2014 είναι το έτος σημαντικών επαιτίων στις ε, σχέσεις Ένωσης και Γεωργίας. Πριν από 10 χρόνια η ε, Γεωργία μπήκε στην, ε, στην πολιτική γυτνίαση και πριν 5 χρόνια έγινε μέλος της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Τέλος να υπογραμμίσω τα πόσα περιμένουμε να επιτύχουμε στην διάσκεψη κορυφής της Ρήγας. Υποσχεθήκαμε να συνεχίσουμε τις ευρύτατες μεταρρυθμίσεις όπως ε, άλλωστε δεσμευτήκαμε και από τη Συμφωνία Σύνδεσης να ε, εδραιώσουμε τη δημοκρατία και να παραμείνουν οι εξελίξεις δημοκρατικές στην περιοχή. Περιμένουμε αρχές του φθινοπόρου να υπογράψουμε τη Συμφωνία Σύνδεσης. Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε σε κοινοτικά προγράμματα όπως είναι το Creative Europe, Horizon 2020, Erasmus και να διερευνήσουμε και νέες οδούς ενεργασίας στην ΕΠΑ, την ΚΕΠΑ. Αρχίζουμε να υλοποιούμε τις διατάξεις Συμφωνίας Σύνδεσης ε, και τη θετική ε, γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιμένω να επιτύχουμε για την άρση θεώρησης διαβατηρίων για σύντομα ταξίδια. Στις μεταφορές, ενέργεια, παιδεία και πολιτισμό επίσης ε, ελπίζουμε να ενισχυθεί ο ρόλος και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχυθεί για την ε, ειρηνική επίλυση των διαφορών. Να έχουμε ισχυρή υποστήριξη και οικονομική από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, συμπεριλαμβανομένων των νέων μέσων συνεργασίας και βοήθειας. Είμαι πεπισμένη ότι μέσω των κοινών προσπαθειών μας θα μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρα σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εξοχοτάτη. Έχουμε πλήθος συναδέλφων που έχουν να κάνουν ερωτήσεις. Κοιτάξτε και το χρόνο. Σας παρακαλώ να περιορίζεστε σε ένα δίλεπτο έκαστος. Ο κύριος Λίσεκ πρώτος, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μίλησε κανείς πολωνικά ως τώρα, θα μιλήσω εγώ. Θα ήθελα, θα ήθελα λέγω, με ακούτε τώρα κυρία Υπουργέ μου. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την αποφασιστικότητα που επέδειξε η γεωργιανή κυβέρνηση στην επίτευξη των στόχων της για τη βελτίωση των σχέσεών μας με την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης. Ξέρετε καλύτερα από μας ότι περιτριγυρίζεστε από χώρες των οποίων η συμπεριφορά δεν είναι σταθερή ούτε της ίδιας ποιότητος. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω κάτι για τα εσωτερικά της γεωργίας. Το μέλλον δηλαδή της, των ανατολικών σας σχέσεων. Η Τι μπορεί δηλαδή να κάνει η Ένωση για να παρέμβει εκτός από τη Μολδαβία και τη Γεωργία και σε άλλες χώρες ώστε να ακολουθήσουν το παράδειγμά σας. Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε την Ουκρανία, το Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Γκόμες. Κύριε, κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστώ που δεχτήκατε να προσέλθετε και να μας κάνετε την παρουσίασή σας. εντυπωσιάστηκα όταν επισκέφτηκα τη χώρα σας σε αντιπροσωπεία πέρυσι του κοινοβουλίου μας και θα ήθελα να σας ρωτήσω πήγαμε και στην Νότια Οσετία όπου ξέρουμε ότι οι Ρώσοι έχουν αρχίσει να χτίζουν το τείχος πώς προχωράνε τα πράγματα Έχετε δει κανένα ξεπάγωμα των σχέσεων. Διότι θα είχε κάτι τέτοιο πολύ θετικά αποτελέσματα στη ζωή των κατοίκων εκεί. Ή μήπως αντίθετα είναι τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα. Υπήρξαν προσδοκίες με την αλλαγή της Προεδρίας ότι τα πράγματα θα μαλάκωναν κάπως. Πέστε μας τι φρονείτε λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Σαλαφράγκας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματο ε, τη ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, θα ήθελα να σα καλωσορίσω, κύριε Υπουργέ. Γνωρίζετε ότι τούτο εδώ το Κοινοβούλιο υποστηρίζει ανέκαθεν και στεναρά ε, την ευρωπαϊκή προσήλωση και προσανατολισμό της χώρας σας και ιδιαίτερα... Εδώ είμαι, εδώ είμαι. και διαστόματος κυρίου Λίσεκ υπόθηκαν αυτά. Ε, Ακούσαμε για μια ημερομηνία για την Συμφωνία Σύνδεσης και ε, είπατε ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες και τα προβλήματα με τη Ρωσία και της εδαφικής ακαιρεότητας που το Κοινοβούλιο αναγνώρισε στο τελευταίο του ψήφισμα που ενέκνε και εν ώψη της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Για τη Συμφωνία Σύνδεσης βλέπετε δυσκολίες να διαγράφονται στον ορίζοντα μετά τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στη Ρωσία. Και ιδιαίτερα ό,τι έχει να κάνει με την εδαφική σας ακεραιότητα, θα ήθελα να ρωτήσω μήπως θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε για τις συζητήσεις που κάνει ο ειδικό εντεταλμένος χώρας σας για τη Ρωσία και ο Ρώσος ε, υφυπουργό Εξωτερικών. Κυρία Υπουργέ, είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Ξέρετε ότι ανησυχούμε για όλο αυτό το θέμα της επιλεκτικής δικαιοσύνης στις χώρες σας. Ο, ε, ο πρώην Πρωθυπουργός καταδικάστηκε σε πενταετία στη φυλάκιση, όπως και ο δήμαρχος της Τυφλίδας ε, κρατείται με περίεργους όρους στις φυλακές. Εγώ δεν προεξοφλώ καθόλου ε, το τεκμήριο της αθότητας ή της ενοχής, αλλά κάπως ε, βλέπουμε ότι υπάρχει μια επιλεκτική δικαιοσύνη και εμποδίζει κάπως την εφαρμογή των θεμελιωδών ελευθεριών και των δικαιωμάτων στη χώρα σας. Τέλος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και να σας ρωτήσω αν μπορείτε να μας δώσετε καμιά λεπτομέρεια των σχέσεων της χώρας σας με άλλες σημαντικές χώρες, Αρμενία, Αζερβαϊτζάν και Τουρκία κυκλοφορούν κάτι φήμες, μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε αυτά που βλέπουμε στον τύπο για ενδεχόμενη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του δικού σας Προέδρου. Ε, επιβεβαιώνονται αυτές. Thank you very much. Ευχαριστώ κύριε Σαλαφράκα. Ο κύριος Φαν Μπάλεν παρακαλώ. Thank you. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που βλέπω την ε, Υπουργό στο Κοινοβούλιο, ήταν και πρέσβης στις κάτω χώρες της χώρας ε, της. συζητήσαμε για πρώτη φορά μαζί όταν είχε εισβάλει στη χώρα σας η Ρωσία και άλλοι συνάδελφοι είχαν ερωτήσει το εξή. Οι Ρώσοι προσπαθούν να διευρύνουν ακόμα και τη ζώνη κατοχής τους βήμα-βήμα. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση τι μπορούμε να κάνουμε ε, και ως Δυτικό Ευρωπαίο, όπως κάνουν και οι Ηνωμένε Πολιτείε για να σας υποστηρίξουμε. Ξέρουμε ότι η παρούσα κυβέρνηση είπε και κατά τη διάρκεια των εκλογών ότι θέλει να γεφυρώσει αυτό το χάσμα με τη Ρωσία, με συνομιλίε. Υπήρξαν συνομιλίες παραγωγικές, ήταν και σε σχέση και με τις άλλες χώρες ανατολική γειτονία προσπαθούν να χαράξουν μία γραμμή. Στην Ουκρανία ξέρουμε τα ίδια προβλήματα υπάρχουν, όπως και στη Γεωργία και στη Μολδαβία τα ίδια. Παντού η Ρωσία θέλει να έχει ε, μια ζώνη επιρροής και βολής της που την ονομάζει μάλιστα και εγγύς πει. Τι είναι αυτά, σε χώρες ανεξάρτητες όπως είστε εσείς και οι γειτονικές σας. Ευχαριστώ ο κύριος Τανζό. Σας ευχαριστώ κύριε Κυρία Υπουργέ. Σας ευχαριστώ για την επίσκεψή σας και για την ε, ε, εισήγησή σας. Δεν θα επανέλθω στις πτυχές που ανέφερε ο συνάδελφος Σαλαφράγκα και που μας ανησυχούν πολύ όσον αφορά την επιλεκτική δικαιοσύνη που φοβόμαστε να αναπτύσσεται στη χώρα σας. Έχω δύο ερωτήματα. Το πρώτο σε σχέση με τη Ρωσία. Ήμουν παρατηρητή στην στιγμή των ε, εκλογών στη Γεωργία που κέρδισε ο Γιώργιν Τρίμ χωρίς ε, καμία αμφισβήτηση. Που κέρδισε η Georgian Dream. Ναι, σχέσει λοιπόν με την ε, Ρωσία υποστήριξαν και φαίνεται πω η κυβέρνηση του κύριου Ιενισβίλη είχε πάλι προσωπικότητε που είχαν τα σε πολύ καλέ θέσει για να γνωρίζουν καλά τη Ρωσία. Όμω σήμερα δεν λειτουργεί το πράγμα, οι Ρώσοι δεν σας κάνουν κανένα δώρο, δεν ε, ε, μπορείτε να επιτύχετε τα όσα είχε επιτύχει η προηγούμενη κυβέρνηση. Βρίσκω αφέλεια να υπάρχει σε αυτήν την προσέγγιση, σίγουρα σε πολιτικό επίπεδο είναι αποτυχία. Δηλαδή σχέση ε, ρύθμισης των σχέσεων με τη Ρωσία δεν έφερε καρπούς. Πώς το εξηγείτε αυτό. Δεύτερη διαφορετική ερώτηση σε σχέση με τις εξωτερικές υποθέσεις της Γεωργίας. Λέγεται πως η Γεωργία θα μπορούσε να είναι σημαντικός ε, συνεισφορέας στην ευρωπαϊκή στρατιωτική επιχείρηση στην Κεντρική Αφρική. Τι γίνεται με αυτό, έχει ήδη αποφασιστεί αυτό και αν ναι, μπορείτε να μας πείτε κάτι περισσότερο. Σας ευχαριστώ. Ο Σερ Γκρέαμ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να χαιρετήσω την παρουσία της Υπουργού Εξωτερικών εδώ και να θυμίσω τη μεγάλη της εμπειρία στις εξωτερικές υποθέσεις ως εκπρόσωπος της χώρας της ε, στο εξωτερικό. Θα ήθελα επίσης να τη συγχαρώ καθώς και την κυβέρνησή της για την ε, τεράστια πρόοδο που έχουν επιτύχει στη Γεωργία. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω για ένα θέμα το οποίο μου ανέφερε συνάδελφοι στην Επιτροπή των Περιφερειών και αφορά την, τον ε, εκλεγμένο δήμαρχο της Τυφλίδας και την ε, αναστολή ε, που έχει πάρει, τη διαθεσιμότητα μάλλον στην οποία έχει τεθεί από τα καθήκοντά του. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο στα γερμανικά. Ευχαριστώ. Περίμενα τον κύριο Μπροκ και του υποσχέθηκα ότι θα απαντήσω στα γερμανικά στις ερωτήσεις. Τώρα αποσιάζει, το πήρα και τηλέφωνο ε, πριν έρθω, είναι καθοδόν για το Βερολίνο. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν μπόρεσα να τον δω, αλλά θέλω να τηρήσω την ε, ε, υπόσχεσή μου και να απαντήσω στα γερμανικά. Ναι, danke Δεν έχετε πρόβλημα. Όχι, λέει ο κύριος Πόσελτ, κανένα. Ωραία. Έχουμε κάτι Γερμανούς εδώ, κανένα δυο στην αίθουσα, λέει ο Πρόεδρος. Και με χαρά θα σας ακούσουν απευθείας. So, ähm, ähm, ich werde dann, ich, ich werde auf... Λοιπόν, ε, ε, θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που είναι αλληλοσυμπληρούμενες και γι' αυτό νομίζω ότι είναι πιο απλό να αναφερθώ σε ορισμένα θέματα, να απαντήσω έτσι κατά θεματικές ενότητες και όχι σε επιμέρους ερωτήσεις, για να επεκταθώ κιόλα. Ποιε είναι οι σχέσεις μας με τους γείτονε και το μέλλον της ε, ανατολικής γειτονία, με ρωτήσατε. Και πώς γίνεται η κατάσταση εκεί με την Ουκρανία, το Αζερβαϊτζάν και την Αρμενία. Ε, με μεγάλη χαρά η Γεωργία εντάχθηκε πριν από πέντε χρόνια στην Ανατολική γειτονία μαζί με άλλες χώρες και τότε πιστέψαμε ότι θα μπορούσαμε από κοινού να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. Δυστυχώς έχουν μείνει δύο ε, χώρες εκτός που ελπίζω τον Αύγουστο να υπογράψουν. Και δυστυχώς είμαστε εμείς μία από τις δύο αυτές χώρες και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Σε ό,τι αφορά τώρα τις υπόλοιπες χώρες, νομίζω ότι είναι κυριαρχικό δικαίωμα κάθε χώρας να αποφασίζει ποιο δρόμο θέλει να επιλέξει. Εξού και δεν πιστεύω εγώ προσωπικά ότι θα πρέπει εμείς να αναμειχθούμε στα εσωτερικά κάποιες χώρες και να προεξοφλήσουμε, να επηρεάσουμε ή να αμφισβητήσουμε ε, κάποιες αποφάσεις συλλημένες από άλλες χώρες. Όλα τα κράτη έχουν διαφορετικές φιλοδοξίες βέβαια στην ε, Ανατολική γειτονία και έχουν τους λόγους τους γιατί το πράττουν. Για την Αρμενία ήταν πολύ ειδικοί λόγοι και προβλήματα που αντιμετώπιζε, θέματα ασφαλείας, θέματα ενεργειακά και εξάρτησης της από τη Ρωσία. Για την Ουκρανία ήταν τελείως διαφορετική κατάσταση. Ελπίζω πάρα πολύ, ανεξαρτήτως των σημερινών τεκτενωμένων στην Ουκρανία, να βρεθεί παρόλα αυτά ένας δρόμος με τη μορφή διαλόγου να λυθεί το πρόβλημα. και πραγματικά ενισχύει ο Ουκρανικός λαός. Σε ό,τι αφορά τη γεωργία δεν υπάρχει κίνδυνος να αλλάξει την απόφασή της η κυβέρνηση, να υπαναχωρήσει και να προσπαθήσει να στρέψει τη χώρα σε διαφορετική κατεύθυνση. Είναι δεδομένη η απόφασή μας. Γνωρίζουμε ότι ο γεωργιανός λαός υποστηρίζει αυτή την πολιτική απόφαση και αυτό είμαι και εγώ βεβαία ότι η Συμφωνία Σύνδεσης θα ε, υπογραφεί τον Αύγουστο. Σε ό,τι αφορά τώρα την πίεση από πλευράς της Ρωσίας και αυτό έχει σχέση και με την υπογραφή ε, της συμφωνία Σύνδεσης. Πιστεύω προσωπικά ότι θα εξακολουθήσει η ρωσική πίεση. Κάνουν φράχτες με σειρματοπλέγματα ακανθώτα, ε, τώρα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων το έχουν σταματήσει λόγω εκεχηρίας. Αλλά μόλις τελειώσουν οι αγώνες πιστεύω ότι θα ενταθεί η εγκατάσταση αυτού του φράχτη και του σειρματοπλέγματος. Ένα δεύτερο που με ανησυχεί ιδιαίτερα είναι η διεύρυνση της ε, λεγόμενης ε, ζώνης ασφαλείας κατά 11 χιλιόμετρα. Το ανέφερα και προηγουμένως στην ομιλία μου. Και υπάρχει φόβος μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες να παραμείνει το σημερινό στάτους κβο. Δηλαδή η Ρωσία που έχει υποσχεθεί να αποσυρθεί και να επαναφέρει τα Ρώσο-Γεωργιανά σύνορα, ε, θα την αθετήσει αυτή την ε, υπόσχεση. Και εμείς φοβούμεθα ότι θα μετατοπίσουν τα σύνορα, κατά 11 χιλιόμετρα έχουν καταπατήσει γεωργιανή επικράτεια. Αυτό είναι πολύ σοβαρό ως πρόκληση και θα πρέπει ε, να το αντιμετωπίσουμε, το θα πάρα πολύ. Και πάλι και ελπίζουμε και προσβλέπουμε στην υποστήριξη των διεθνών οργανισμών και των εταίρων μας, καθώς επίσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια προσβλέπουμε και στην υποστήριξη του Κοινοβουλίου σας. Για τα οδοφράγματα στην Νότια Οσετία που ε, χωρίζουν ε, την επικράτεια εκεί από εκείνη την επικράτεια που είναι υπό τον έλεγχο της γεωργιανής κυβέρνησης δυσκολεύουν πάρα πολύ τη ζωή των ανθρώπων. Τα θεμελιώδη τους δικαιώματα παραβιάζονται, τα ουσιαστικά τους δεν έχουν καμία δυνατότητα ούτε να μετακινούνται ελεύθερα, ούτε να μιλούν καν τη μητρική τους γλώσσα στο σχολείο. Ε, δεν έχουν μάθημα στα Γεωργιανά δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε άλλες δομές κοινωνικές υγείας, σε υπηρεσίες υγείας ή πρόνοια και οι οικογένειες που πλήττονται από αυτή την κατάσταση βεβαίως ε, υποφέρουν πάρα πολλά δεινά. Κύριε ρωτήσατε ε, αν οι καταστάσεις είναι ε, το εξίσου ψυχρές όπως και στο παρελθόν δυστυχώς δεν έχουμε εντατικές σχέσεις με τον πληθυσμό ε, πέρα από τη γραμμή κατοχής. Προσπαθούμε να έχουμε επαφές, προσπαθούμε έτσι να δείξουμε όσο μπορούμε και να βοηθούμε όσο μπορούμε ε, το κόσμο εκεί. Υπάρχουν διάφορα και κοινωνικά προγράμματα, προγράμματα στον τομέα της υγείας και ο πληθυσμός από την άλλη πλευρά της ε, διαχωριστικής γραμμής μπορεί να υποφελείται εάν επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτά τα προγράμματα. Έχουμε την επιθυμία πραγματικά ο κόσμος να συμμετέχει και να δείχνουμε ότι είμαστε πρόθυμοι πάντα να βοηθούμε. Γιατί αυτή η διαχωριστική γραμμή δεν είναι κάτι που μπορούμε να δεχθούμε εμείς. Είναι κατοχή και είναι κάτι που έχει υψώσει ο κατακτητής κατά του λαού. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Ιβανισβίλη, ε, είχε ε, δημιουργήσει ένα είδος διαλόγου με ένα ειδικό εντεταλμένο. Κατά τα άλλα πρέπει να σας πω η κυβέρνηση παραμένει η ίδια, μόνο ο Πρωθυπουργό έχει αλλάξει. Έχει επαφές με τον ε, αντι... Ε, συγγνώμη, υφυπουργό εξωτερικών της Ρωσίας γίνονται τακτικές επαφές και έτσι μπορούν και πάλι να εξάγονται γεωργιανά αγροτικά προϊόντα προς τη Ρωσία. Αλλά μέχρι εκεί η συνεργασία νομίζω, ε, σε αυτή τη δεύτερη φάση των σχέσεων με τη Ρωσία. Αυτό ήταν το επίτευγμα. Βεβαίως η Γενέβη παραμένει ε, πιο σημαντική ε, πόλη για το διάλογο ε, Ρωσίας-Γεωργίας, αλλά δυστυχώς δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος σε αυτό τον τύπο των συνομιλιών. Μετά από 26 γύρους η κατάσταση παραμένει όσοι είχε στην αρχή το 2008. Τώρα ελπίδα έχουμε ότι τα νέα δεδομένα, για παράδειγμα, ελπίζω πάρα πολύ να ολοκληρωθούν με επιτυχία Ολυμπιακοί Αγώνες στο Σότσι και με αυτά, ε, μετά το θετικό αυτό, πώς να το πω, κλίμα ε, και το θετικό γεγονός για τη Ρωσία να βοηθήσει κάπως και να επηρεάσει και τις συνομιλίες της Γενέβης με τρόπο θετικό όσο γίνεται. Εκτός αυτού, υπάρχει και κάτι άλλο στη Γενέβη. Έχουν μπει κάποιοι νέοι παράγοντες εκεί η Ελβετία που προεδρεύει αυτό τον καιρό στον ΟΑΣΕ. Προσεχώς θα έχουμε και ένα νέο ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφέρειά μας και με αυτά τα νέα πρόσωπα που να συμμετέχουν στο διάλογο στη Γενέβη μπορεί ενδεχομένως να κινηθούν τα πράγματα ε, για να αποτελματοθούν. Ακούστηκε κάτι για ενδεχόμενη συνάντηση του Προέδρου της ε, Δημοκρατίας Γεωργίας με τον Ρώσο Πρόεδρο. Αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ επίκαιρο και καυτό στη συζήτηση στη χώρα μου. Ένας δημοσιογράφος σε μια συνέντευξη που ρώτησε τον Ρώσο Πρόεδρο εάν θα ήταν πρόθυμος να συναντήσει τον Γεωργιανό ομολογό του. Και η απάντηση ήταν καταφατική. Οπότε το θέμα στη Γεωργία έπαιξε πάρα πολύ ψηλά και έγινε πάρα πολύ επίκαιρο, το πήραν ε, όλοι οι δημοσιογράφοι και το κυκλοφόρησαν. Δεν υπάρχει όμως προετοιμασία αυτή τη στιγμή για μια τέτοια συνάντηση. Έχει μείνει σε αυτή τη μία απάντηση του Προέδρου Πούτιν ε, σε συνέντευξη τύπου. Ούτε έχουν κάνει οι Ρώσοι κανένα βήμα για να ζητήσουν ε, συνάντηση στο ψηλότερο επίπεδο μεταξύ των εκπροσώπων των κρατών αυτών. Στις 5 Μαρτίου προβλέπεται η νέα συνάντηση Αμπασίτσε Καράσιν και ακούμε από ρεσικής πλευράς ότι θα συζητηθεί και ε, αυτό το θέμα. Θα το θέσει ο Ρώσος δηλαδή το θέμα της συνάντησης των Πρόεδρων. Προετοιμασία δεν γίνεται αυτό τον καιρό, αλλά δεν αποκλείουμε και τίποτα. Τουλάχιστον εμείς έχουμε προθυμία, εφόσον ζητηθεί ή οργανωθεί τέτοια συνάντηση, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά που να έχει και συγκεκριμένα αποτελέσματα, όχι μια συνάντηση για να γίνει, τότε θα ε, φροντίσουμε και εμείς και είμαστε βεβαίως υπέρ του να διεξαχθεί και να λάβει χώρο. Με ρωτήσατε εάν η κυβέρνηση επιδεικνύει κάποια αφέλεια όταν πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο του διαλόγου και με άλλα μέσα μπορεί κανείς να βελτιώσει τις σχέσεις του με τη Ρωσία. Και μήπως θα αποτύχουν όλες αυτές οι απόπειρες, οι προσπάθειες που κάνει η γεωργιανή κυβέρνηση. Κοιτάξτε, πρόσφατα συνεδρίασε η Επιτροπή ΝΑΤΟ Γεωργίας εδώ στις Βρυξέλλες και πολλοί εκπρόσωποι των χωρών μελών του ΝΑΤΟ μας ευχαρίστησαν ρητά πραγματικά για τα επικοδομητικά βήματα που κάναμε προς την κατεύθυνση της Ρωσίας και προσπαθούμε όσο γίνεται να αποκλιμακώσουμε την ένταση και να τη κρατήσουμε σε χαμηλά επίπεδα. Αυτό είναι καλή προϋπόθεση και για τους εταίρους μας και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τον ΝΑΤΟ. Το θέμα Γεωργία-Ρωσία να το συζητάμε με νυφαλιότητα και ηρεμία. Αν μας ρωτάτε τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να συνεισφέρει προς την κατεύθυνση αυτή, να χαλαρώσει πίεση, θα πρέπει να στείλετε ένα σαφές μήνυμα ότι δεν μπορεί καμία τρίτη χώρα να επηρεάσει τις αποφάσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ε, μια άλλη χώρας να ενταχθεί στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν σταλεί αυτό το σαφές μήνυμα, θα βοηθούσε. Και δεν μπορεί μια τέτοια εμπεραλιστική λογική που ε, έχει μόσχα να αποτελέσει εμπόδιο και τροχοπέδι. Αν στείλετε αυτό το μήνυμα θα χαλαρώσει η πίεση, θα καταλάβει η Ρωσία ότι η Γεωργία θα πρέπει ανεξάρτητα από τη ζώνη επιρροής και τη Ρωσία να μπορεί να αποφασίσει που έχει αποφασίσει το μέλλον της και θα ακολουθήσει αυτή την κατεύθυνση ό,τι και να γίνει. Το ίδιο ισχύει και για το ΝΑΤΟ. Ένα σαφέ μήνυμα προς τη Ρωσία πρέπει να σταλεί ότι δεν έχει δικαίωμα βέτο η Ρωσία για το ΝΑΤΟ, για την απόφαση ε, του ΝΑΤΟ. Αυτό μπορεί να βοηθήσει να ε, σταθεροποιηθεί η κατάσταση και να καταλάβουν όλοι ε, ότι κανείς δεν μπορεί να απειλήσει αυτές τις προτεραιότητες της γεωργιανής εξωτερικής πολιτικής. Επίσης πιστεύω ότι και για τους ανθρώπους που ζουν στις κατεχόμενες περιοχές Στο συγγνώμη. Αυτό είναι καιρό στέι στη Γεωργία όμω όχι στι Βρυξέλλε. Δεν κρύος εδώ. Το είδαμε. Στο Σότσι δεν έχει χιόνι. Εσείς που κρυώσατε. Chairman, I think the foreign minister needs a glass of your special palinka. Πρόεδρε, λέει ο κύριος Γότσον, ε, ε, υπουργός ε, χρειάζεται ένα ποτηράκι από την ειδική παλίνκα που έχετε, το δικό σας το ποτό, πρόεδρε. Καλά, άτυπη ήταν αυτή η πρόταση. Λοιπόν, επανέρχομαι για την επιλεκτική δικαιοσύνη που με ρωτήσατε είπατε ότι συνελήφθη ο δήμαρχος της Τυφλίδος. Αυτό δεν ισχύει φυσικά. Και ο πρώην πρωθυπουργός της Γεωργίας σήμερα, το έμαθα εδώ σήμερα, καταδικάστηκε σε πενταετή φυλάκιση. Θα ήθελα να πω το εξή μόνο. Αυτή η φάση πιστεύω έχει ε, παρέλθει η επιλεκτική δικαιοσύνη. Έχουμε δείξει κατά τη διάρκεια του έτους ότι η γεωργιανή δικαιοσύνη είναι πλέον ανεξάρτητη, πιο ανεξάρτητη από ποτέ και από μακριά από μένα η αντίληψη ότι ε, η γεωργιανή δικαιοσύνη είναι 100% ανεξάρτητη και δεν δέχεται καμία ε, επιρροή από πουθενά και από κανένα. Δεν λέγω κάτι τέτοιο, αλλά αν συγκρίνουμε την κατάσταση με αυτή που επικρατούσε πριν από χρόνια, είναι η διαφορά αισθητή. Είναι επίσης σαφές ότι και στη Γεωργία ουδής είναι υπεράνω του νόμου. Και όταν μια δίκη γίνεται με διαφάνεια, με στοιχεία πάντα και ε, αποδείξεις, τότε δεν θα πρέπει κανείς να εκφράζει ούτε μία κριτική ούτε να αναφέρεται σε επιλεκτική δικαιοσύνη στη Γεωργία. Διότι σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις ε, η εισαγγελία κατέθεσε αδιάσυστα αποδεικτικά στοιχεία και ε, το ανεξάρτητο δικαστήριο που είναι πιο ανεξάρτητο από ό,τι στο παρελθόν και που ουδέποτε επαναλαμβάνω ήταν τόσο ανεξάρτητη δικαιοσύνη όσο σήμερα κατέληξε σε μία απόφαση. Πριν από μερικά χρόνια κάτι τέτοιο θα ήταν τελείως αδύνατο. Επίσης, ο πρώην Πρωθυπουργό αναγνωρίστηκε ένοχος για τρία δικήματα και στο παρελθόν θα είχε καταδικαστεί για περισσότερα χρόνια διότι υπήρχε ε, άθροισμα των ποινών. Ε, η νυν κυβέρνηση το έχει καταργήσει αυτό και τιμωρείται απλώς με την ποινή που επιβάλλεται για το σοβαρότερο αδίκημα και όχι με 15-20 χρόνια που θα ήταν η ποινή του στο παρελθόν, αθρηστική δηλαδή και πολύ πρόσφατα μέχρι πριν από 2 και 3 χρόνια. Ε, όσο δε για τον δήμαρχο Τυφλίδος, δεν κρατείται στη φυλακή. Ε, διεξάγονται έρευνες ακόμα και πριν ολοκληρωθούν, νομίζω δεν θα έπρεπε να ε, έχουμε προεξοφλήσει τίποτα. Οι δίκες επίσης παρακολουθούνται και από τον ΟΑΣΕ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις πιο πρόσφατες εκθέσεις του ΟΑΣΕ και της Ένωσης γίνεται λόγος για την ανεξάρτητη πλέον δικαιοσύνη και τα ανεξάρτητα δικαστήρια στη Γεωργία και για τις δίκες και διαφανείς δίκες. Νομίζω αυτό είναι επίτευγμα των τελευταίων ετών. Όπου καταδικάστηκαν 300.000 άνθρωποι στη Γεωργία και πάρα πολλοί αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση. Πλέον δεν ισχύει κάτι τέτοιο και είναι κάτι το οποίο χαροποιεί πάρα πολύ τον κόσμο στη Γεωργία και μάλιστα τον καθιστά και πάρα πολύ περήφανο το λαό μας. σε λίγο καιρό θα έχουμε δημοτικές εκλογές, δεν το είπα καθόλου στην πρώτη ομιλία μου αυτό, και ε, είναι στο προπαρασκευαστικό στάδιο. Άκουσα σήμερα ότι η μισή ότι θα υπάρχει το όριο του 50% για να εκλεγεί ένας δήμαρχος. Δηλαδή πρέπει να έχει απόλυτη πλειοψηφία. Και δεν εκλέγεται μόνο ο δήμαρχος στη Διφλίδα, αλλά και σε 12 άλλες πόλεις ε, και η τοπική κυβέρνηση. Δηλαδή και αυτό είναι ένα βήμα προς τη δημοκρατία και παρακολουθούμε και ε, σεβόμαστε πάρα πολύ τις συστάσεις που έχουμε λάβει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από άλλους εμπειρογνώμονες και πιστεύω ότι με τις δημοτικές εκλογές θα μπορέσουμε να δώσουμε και τις τελευταίες εξετάσεις για τη δημοκρατία στη Γεωργία και να δούμε κατά πόσο απειλείται ή δεν απειλείται. Και δεν θα πρέπει να ξαναπαντήσω σε άλλη ερώτηση για το αν απειλείται η δημοκρατία στη Γεωργία. Νομίζω ότι απάντησα πάνω κάτω στις ερωτήσεις σας. Α, για την Αρμενία, Αζερπαϊτζάν και την Τουρκία κάτι με ρωτήσατε και με τις τρεις αυτές χώρες έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Με το Αζερμπαϊτζάν και την Τουρκία βεβαίως πιο εντατικές από ό,τι με την Αρμενία. Γιατί έχουμε δεσμούς ε, οικονομικούς και πολλά ενεργειακά προγράμματα, αλλά η Γεωργία και η Τυφλίδα είναι ένα σημείο που μπορούν να συναντηθούν όλοι από την περιοχή μας και να υπάρξει συνεργασία μεταξύ όλων των χωρών της περιοχής. Το Αζερβαϊτζάν και η Τουρκία είναι σημαντική εμπορική μας εταίροι και το πιο πρόσφατο ε, έργο είναι μια σιδηροδρομική γραμμή Μπακού Τυφλίδα Κάρς που θα εγκαινιαστεί το 2015 Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα ακόμα παράδειγμα της περιφερειακής μας συνεργασίας. Ja, ich glaube, das war's auch. Νομίζω ότι η απάντηση. Thank you very much. Σας... What, uh, former... Θυμάμαι ότι ένας πρώην πρόεδρος της Μακεδονίας έλεγε για τα Βαλκάνια ότι και η μνήμη και τα μαχαίρια είναι πολύ μακρά. Ποιες νύχτες. Ρε. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Η χώρα σας θα παραμείνει ελπίζω στο δρόμο προς την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή ανακλήρωση. <coughs> Κυρίε και κύριοι σα καλησπερίζω. Μου ζητήσανε να προεδρεύσω στις ψηφοφορίες. Εάν λοιπόν συμφωνείτε σε λίγο θα αρχίσουμε. Πρέπει όμως να δείξετε κατανόηση γιατί για πρώτη φορά στη ζωή μου προεδρεύω. Να είστε λοιπόν υπομονητικοί, θα αρχίσουμε ζητώντας, ρωτώντας τον εισηγητή αν θέλει να κάνει καμία εισηγησούλα του θέματος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, όχι δεν χρειάζεται να επανέλθω στο κείμενο, ευχαριστώ απλώς τους συντονιστές και τους κοιόδης με τους οποίους συνεργαστήκαμε πολύ καλά. Δύο θέματα μόνο Πρώτον, υπάρχουν μερικές τροπολογίες επί τους οποίων, ζήτησα καταψήφιση όχι ως προς την ουσία αλλά γιατί νομίζω ότι ε, τυπικά ε, επιβαρύνουν το κείμενο. Αν και πολλές από αυτές είναι πολύ σωστές. Βέβαια όταν ζητάμε σφαιρική αντιμετώπιση σημαίνει ότι εξ ορισμού μπορούμε να μιλήσουμε για όλα, αλλά αν μιλήσουμε για όλα μετά νερώνεται το θέμα. Και δεύτερον, πολύ συγκεκριμένο, η τροπολογία 90 που κατέθεσε η κυρία Κρόνμπεργκ για την παράγραφο 16. Στην παράγραφο 16 ίσως μια υπερβολική επίκριση για το συντονισμό του σχεδιασμού της εξωτερικής πολιτικής μεταξύ των διαφόρων παραγόντων της. Η κυρία Κρόνμπεργκ κατέθεσε μια τροπολογία που αφορά όμως την εφαρμογή. Εγώ μίλησα για το σχεδιασμό εκείνη για την εφαρμογή. Είναι μεν συμπληρωματικά αλλά δεν είναι τα ίδια. Γι' αυτό λέω να κρατήσουμε την αρχική παράγραφο που είναι επικριτική για το σχεδιασμό και να προσθέσουμε προφορική τροπολογία με προφορική τροπολογία το μεγαλύτερο τμήμα του κειμένου της κυρίας Κρόνμπεργκ ως προσθήκη. Έτσι θα έχουμε μία προφορική τροποποίηση για την παράγραφο 16. Διαβάζω αγγλικά. Μετά από το policies on the ground να λέει takes note και τα λοιπά. Μέχρι εκεί που λέει CFSP activities. Αυτό προτείνω λοιπόν. Αυτή είναι η πρότασή μου. Ωραία, όταν θα φτάσουμε στην 50 θα το ξαναπούμε αυτό. Λοιπόν, και τώρα στη γλώσσα του Σέξπιρ. Να αρχίσουμε you have, uh, amendment Τροπολογία 4. Υπέρ. Thank you. Who votes again? Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πέντε. υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 5. εγκρίνεται, εγκρίνεται. Έξι. Υπέρ κατά αποχές απαρρίπτεται. Συμβιβαστική ένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται εννέα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δώδεκα είναι μάλιστα του κυρίου Βαν Όρντεν. Δώδεκα. Υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απαρρίπτεται. Συμβιβαστική Δύο υπέρ. Κατά. Χες εγκρίνεται. Συμβιβαστική τρία υπέρ κατά ποιες εγκρίνεται εννέα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά χες απορρίπτεται 21 υπέρ 21 υπέρ υπέρ κατά χες εγκρίνεται 22 υπέρ ε, κατά κατά χες κρίνεται 23 υπέρ κατά χες παρύπτεται συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά βόχες νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά θα επαληθεύσω ηλεκτρονικός την 29 έληξε εγκρίνεται Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Χες εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Χες εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές γκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές απαρρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, όχι, απορρίπτεται, με συγχωρείτε. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Χες εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά. Χες εγκρίνεται. 46, όχι, όχι 46, 42. 42 υπέρ, υπέρ, κατά. Ποιες απορρίπτεται 46 υπέρ, κατά. πρέπει να γυρίσουμε πίσω στη 43 πρώτα, 43 γιατί δεν κατέπεσε επειδή κατε, ε, απερίφθη η 42. Λοιπόν, ποιος είναι υπέρ της 43, υπέρ, θα, θα, πόχες, επαλήθευση, επαλήθευση, 43. Έληξε. Εγκρίνεται. Με μία ψήφο διαφορά. Μάλιστα. Είπαμε ήταν 43. Ξανά. Ξανά ψήφισαν όλοι. Ε, έληξε. Τώρα απορρίπτεται με δύο ψήφους διαφορά. 46 τώρα. 46. Όχι. 45. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω τα ίδια με πριν, ε. Επαλήθευση τη 45. Επαλήθευση τη 45. Έληξε τα ίδια. 13 υπέρ, 15 κατά. Απορρίπτεται. 44. 44 υπέρ, κατά, οχες, απαρρίπτεται. 46 υπέρ κατά επαλήθευση 46 επαλήθευση 6 επαλήθευση ψήφισατε όλοι ένας ακόμα ένας ακόμα Κάποιος ξέχασε να ψηφίσει κάποιος. Α, εντάξει τώρα. Τα ίδια, 13-15. Απορρίπτεται. 47 υπέρ. Α. Σαράντα επαλήθευση. Σαράντα επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι, ναι. Έληξε 16 υπέρ 12 κατά, εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Yes, εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Yes, εγκρίνεται. 50 τώρα, 50 ο κύριος Ντανζό μας προτείνει προφορική τροποποίηση, την προσθήκη δηλαδή του κειμένου της κυρίας Κρόνμπεργκ. Ναι, εντάξει, συμφωνούμε. Η 50 με την τροποποίηση, λοιπόν, υπέρ. Όπως πρότεινε ο κύριος Ντανζάν, υπέρ. Κατά. Yes εγκρίνεται 51 υπέρ κατά πόχες εγκρίνεται 52 υπέρ κατά πόχες απορρίπτεται αλλά ας επαληθεύσουμε 52 επαλήθευση 13 υπέρ 15 κατά απορρίπτεται. 53 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται αλλά θέλω να επαληθεύσω την 60 ναι απορρίπτεται 61 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 62 υπέρ κατά ποιες παρύπτεται 63 υπέρ κατά ποιες εγκρίνεται αλλά να επαληθεύσουμε την 63 63 ηλεκτρονικά. Όλοι παρακαλώ ε, και όλες. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται με ευρεία πλειοψηφία. Δεν ήταν όμως τόσα πολλά χέρια ψηλά, τέλο πάντων. 66 υπέρ κατά χες απορρίπτεται. 64 υπέρ κατά χες μπορείπτεται 65 υπέρ της 65 κατά χες μπορείπτεται 67 υπέρ κατά χες 67 επαλήθευση. 67 επαλήθευση. Ισοψηφία απορρίπτεται. 68 υπέρ της 68 κατά Επαλήθευση. 68. Επαλήθευση. Πάλι ισοψηφία, πάλι απορρίπτεται. 69. Υπέρ. Α. Yes. Εγκρίνεται. 70 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση. Εγκρίνεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίπτεται 72 υπέρ κατά χες απορρίπτεται 73 υπέρ κατά χες απορρίπτεται 74 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 76 υπέρ κατά συγκρίνεται εγκρίνεται 77 πίπτη, 3 υπέρ κατά ποιες εγκρίνεται δύο υπέρ κατά αεπαλήθευση ηλεκτρονικά um, εγκρίνεται με διαφορά μιας ψήφου Τώρα οι γνωμοδοτήσεις από την ΑΝΑΠΤ για να δω, για να δω εδώ Δεν μπορούμε όλες μαζί. Δεν μπορούμε. Λοιπόν, Ανάπτ 1 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Ανάπτ 2 υπέρ κατά εποχέ εγκρίνεται. Ανάπτ 3 υπέρ κατά Α, όχι, επαλήθευση, επαλήθευση για την ΑΝΑΠΤ 3. Λήθευση εγκρίνεται. Ανάπτ 4 υπέρ κατά αποχές πορύπτεται ανάπτ πέντε, υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται ανάπτ έξι, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ανάπτευτα υπέρ κατά χες εγκρίνεται ανάπτωχτο υπέρ κατά χες εγκρίνεται ανάπτενέα υπέρ κατά χες εγκρίνεται. Τώρα η γνωμοδότηση από την Επιτροπή Γυναικών Συμβιβαστική 9 9 Συμβιβαστική 9 η γνωμοδότηση από την Επιτροπή Γυναικών η προτείνει το συμβιβαστική 9 υπέρ κατά μα πως τολμάτε αποχές εγκρίνεται και επομένως όλες οι άλλες καταπίπτουν και τώρα η τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά ο Άρχεται η ψηφοφορία. Δύο ακόμα, ψηφίστε, ψηφίστε, εντάξει τώρα, εντάξει. Εγκρίνεται 23 ψήφοι υπέρ, μία κατά και πέντε αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Okay, uh, dear colleagues. Uh, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να συνεχίσουμε. Έχουμε και άλλα θέματα. Και επίσης έχουμε μόλις ένα τέταρτο για το επόμενο θέμα μας. Το οποίο είναι η σύναψη της τροποποίησης της στόχα στο πρωτόκολλο του Κιώτου στη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή και την από κοινού εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων. Η συγκητής είναι ο κύριος Τάραντ των Πρασίνων και Ελεύθερης Ευρωπαϊκής Συμμαχίας. Θέλει να πει τίποτα ο συγκητής. Και έχουμε και για τη γνωμοδότηση κάποιον ε, ε, αρμόδιο, αλλά πρώτα ο εισηγητής. Ευχαριστώ. Εισαγωγή λέτε να κάνω. Τη μακρά εκδοχή. Γιατί υπάρχει και η σύντομη που λέει να υποστηρίξουμε την ε, έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος γιατί λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία και όλες τις διασκέψεις που είχαμε και εμείς στο Κοινοβούλιο και οι άλλοι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική αλλαγή και την πολιτική μας. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω περισσότερα. Αυτά αρκούν. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Άλλος κανείς θέλει το λόγο για το θέμα αυτό. Α, ο κύριος Χάουιτ. Σκιώδη των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Παρακαλώ. Δεν θα μιλήσω περισσότερο από τις ηγητής. Απλώς ήθελα να μιλήσω για τη σύσταση. Τη βρίσκω κάπως παράξενο. Γιατί στη χώρα μου γίνεται δημοσία συζήτηση για τις κλιματικές αλλαγές και να έρχομαι εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο μετά Υποστηρίζουμε αυτή την τροποποίηση στο πρωτόκολλο του Κιώτο γιατί η ε, η περιβαλλοντική διπλωματία είναι σημαντικό κομμάτι της δικής μας δουλειάς γιατί χώρες που θέλουν να συνυπογράψουν και να είναι στατηγική μας θέση όπως η Ρωσία και η Κίνα θα πρέπει να τηρήσουν το πρωτόκολλο αυτό και Μέχρι ότου γίνει και το Κιώτο 2 θα υπογραμμίσουμε έτσι τον ηγετικό ρόλο της Ένωσης για τα θέματα του περιβάλλοντος. Ε, παρατείνεται η περίοδος των δεσμεύσεων και ελπίζουμε πως έτσι θα, υπάρξει, θα είναι επιτυχής και η επόμενη συμφωνία του Κιώτο. Για όλους αυτούς τους λόγους υποστηρίζω λοιπόν την συνυπογραφή της τροποποίησης. Σας ευχαριστώ κύριε Βότσον. Γιατί οι άλλοι σκιώδεις δεν θέλουν τον λόγο, οπότε μπορείτε να μιλήσετε. Ναι, θέλω να συμφωνήσω με τον εισηγητή ότι η κλιματική διπλωματία πρέπει να αποτελέσει ένα απόστατο τμήμα της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης και η δέσμευση στην συμφωνία της ΔΟΧΑ θα πρέπει να είναι προτεραιότητα και να θίγεται, να αναφέρεται κατά προτεραιότητα στις διμερείς επαφές. Ε, υπάρχει σύγκληση των απόψεων των επιστημών όσον αφορά τους κινδύνους και τη ζημιά που ήδη έχει προκληθεί στα καιρικά ε, φαινόμενα και ε, γι' αυτό και θα πρέπει να προχωρήσουμε στην σύναψη αυτής της τροποποίησης. Κάποιος άλλος θα ήθελε το λόγο. No. If not, then I... Εφόσον όχι, κλείνουμε τη συζήτηση για τώρα και θα πρέπει να ψηφίσουμε στην ε, ΕΠΕΞ στις 23 Μαρτίου. Στις 3 Μαρτίου, με συγχωρείτε και μετά να στείλουμε την ε, δική μας ε, γνωμοδότηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος που ψηφίζει τις 6 και η ψηφοφορία στην Ορομέλεια θα πρέπει να γίνει τον Απρίλιο. Θέλει κάποιος από την Κομισιόν να πάρει το λόγο. Όχι, ευχαριστώ πολύ λοιπόν και μπορούμε έτσι να κλείσουμε αυτό το θέμα. Mm. Uh, I can suspend. Λοιπόν, και τώρα θα σταματήσουμε τη συνεδρίασή μας μέχρι τις 6 παρατέταρτο, οπότε και θα γίνει μια ε, σύσκεψη μαζί με την αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ισλανδία και την ε, Νορβηγία και την Ελβετία καθώς και τη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, που θα αφορά τις επιπτώσεις του ελβετικού δημοψηφίσματος και η σε αυτή θα είναι και κλεισμένων των θύρων. Οπότε σας ευχαριστώ και διακόπτουμε για 10 λεπτά.